Äh, λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε αλλάξει λιγάκι την ημερήσια διάταξη. Ελπίζω να είσαστε σύμφωνοι με τις αλλαγές αυτές. Να σας πω ότι έχουμε σήμερα διερμηνία σε πολλές γλώσσες. Η συνεδρία μας επίσης ε, ε, βρίσκεται και είναι και online. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Όχι. Οπότε εγκρίνονται και αυτά. Πάμε στο θέμα της απαλλαγής για τους διάφορους φορείς. Πάμε λοιπόν δηλαδή στα σημεία 9, 10 και 11 που τα έχουμε φέρει πιο μπροστά στη σειρά στην ημερήσια διάταξη να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια για να μας ε, πει πώς θα προχωρήσουμε. Έχουμε μια έκθεση που έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και βεβαίως να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στην ε, εισηγήτρια τη Μόνικα Μακοβέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την ψηφοφορία του Μαΐου, σε συνεργασία με τους συντονιστές, αποφασίστηκε να θεωρήσουμε ως βάση για το δεύτερο σχέδιο έκθεσης τις εκθέσεις που εγκρίθηκαν στις 10 Μαΐου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και το επόμενο βήμα πά τη διαδικασίας είναι η κατάθεση τροπολογιών. προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου. Αλλά όπως ε, έγραψα και στα προηγούμενα μηνύματα που σας έστειλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους συναδέλφους, εγώ θα στείλω ε, σχέδιο των αλλαγών σε όλους δύο-τρεις μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, ώστε να δείτε λίγο ποιες είναι οι προθέσεις μου και να αποφύγουμε επανάληψη τροπολογιών από ε, τους συναδέλφους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται χρόνο προκειμένου να βελτιώσουν ή να αρχίσουν να εφαρμόζουν κάποια από τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία οδήγησαν στην αναβολή της απαλλαγής τους και επομένω είναι προς το συμφέρον και των οργανισμών αυτών να έχουν αρκετό χρόνο ε, για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και επιλέξαμε αυτή την άγουσα. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι θα γίνει η συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών στις 5 Σεπτεμβρίου πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, αλλά όπως σας είπα θα έχετε λάβει ήδη στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου τις δικές μου τροπολογίες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι είμαι σε στενή επαφή και με τις τρεις αρχές. Συζήτησα με τους διευθυντές ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων και για το, του Οργανισμού Φαρμάκων. Ε, ε, δόθηκαν κάποιες οδηγίες για μέτρα τα οποία μπορούν να λάβουν για να αποφύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων χρησιμοποιώντας Ω πηγή τι κατευθυντήρε γραμμές του ΟΣΑ για τις σύγκρουση συμφερόντων και για την ε, αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, για παράδειγμα, ζητήθηκε έκθεση από την ίδια την αρχή για το πώς μπορεί να διασφαλίσει ανεξαρτησία του επιστημονικού έργου, ανεξαρτησία από τον ε, κλάδο και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για σχετικά ζητήματα. Διαπιστώνω ότι ε, δεσμεύονται και θέλουν ε, να ε, υλοποιήσουν όλα αυτά τα μέτρα. Βέβαια γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν αμέσω όλα τα μέτρα, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον η εφαρμογή κάποιων και η δέσμευση που αναλαμβάνουν κατ' εμέ είναι ικανοποιητική και θα ήμουν διατεθειμένη από εκεί και πέρα να τους παραχωρήσουν απαλλαγή. Ε, όπως συζήτησα με τις διάφορες αρχές, θα μας στείλουν τα τελευταία τους αποτελέσματα στα μέσα Αυγούστου περίπου και αν θέλετε φυσικά μπορώ να τα διαβιβάσω σε όλους από εκεί και πέρα όταν θα τα λάβω από τις αρχές. Συζήτησα επίσης με τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλέων για την περίπτωση της αρχής ε, περιβάλλοντος και την αρχή των, ε, οργανισμών φαρμάκων και ε, με την αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων δεν συνομίλησε, διότι όπω γνωρίζετε, ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου παρετήθηκε ακριβώ για λόγου σύγκρουση συμφερόντων. Ε, συζήτησα λοιπόν ε, με τον εκτελεστικό διευθυντή κάποια στοιχεία τα οποία συζήτησα μαζί του ε, βρίσκονται στα έγγραφα τα οποία έδωσα και στις ίδιες τις αρχές και μίλησα και με τον Επίτροπο Ποτέτσνικ που είναι αρμόδιος για την αρχή περιβάλλοντος. Εν τω μεταξύ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβα ένα έγγραφο με ένα πρόγραμμα δράσης μια κάποιας μορφής για το τι ζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Περιβάλλοντος. Ε, σήμερα έλαβα και ένα mail από το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά θα συνεχίσω την αλληλογραφία μαζί τους για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς, εγώ δηλαδή και οι υπηρεσίες, ε, συνεργαζόμαστε επί του ζητήματος αυτού και σας διαβεβαιώ ότι η πρόθεσή μου είναι να υποστηρίξω τις ε, τρεις αρχές, να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα εάν δεν μπορέσουν ε, να κάνουν να λάβουν μέτρα ώστε να επιληθούν όλα τα προβλήματα μέχρι τέλη Αυγούστου τότε θα παρακολουθήσουμε τα ζητήματα αυτά και στις εκθέσεις και στα επόμενα έτη, από κοινού φυσικά και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για κάποια από τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ε, φαντάζομαι ότι αρκετοί θα θέλουν το λόγο για το θέμα. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Βράτω με τις ευκαιρίες για να σχολιάσω κι εγώ κάποια πράγματα σε σχέση με την απαλλαγή. Καταρχάς η διαδικασία της ε, απαλλαγής είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το Κοινοβούλιο και αυτό το εργαλείο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με απόλυτη ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε επακριβώς τα επιχειρήματα και νομίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχων του Προπολογισμού ε, σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτούς τους ευρωπαϊκούς φορείς ε, κοίταξε πολύ προσεκτικά τις περιπτώσεις. Προφανώς υπήρχαν διάφορες ε, αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των, ε, των ομάδων. Κάποιοι είπαν ότι πρέπει να παραταθεί λίγο η διαδικασία, κάποιοι είπαν ότι δεν επαρκούν τα, τα ε, επιχειρήματα για να ζητηθεί ή να προταθεί η απαλλαγή. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική διαδικασία, αλλά η ολομέλεια του Κοινοβουλίου και προφανώς το ανώτατο όργανο λήψη απόφασης εδώ ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία τις εκθέσεις Μακοβέη, οπότε με βάση αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε. Βεβαίω έγιναν και άλλε συζητήσει, έγινε και ανταλλαγή επιστολών για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πω ότι ο πρόεδρος, ο Μαρτίν Σούλτ έκανε κάποιε συζητήσει μαζί μου ώστε σε σχέση με το θέμα αυτό, αλλά και για τις δύο ακροάσεις που θέλουμε να κάνουμε, ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ε, έχει το καθήκον να μελετήσει τις ε, περιπτώσεις αυτές και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως δεν θα γίνει κατά αναγκή εδώ για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον έτσι ώστε να φροντίσουμε ότι η άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού θα συνεχίσει να έχει την ίδια βαρύτητα ούτως ή άλλως οι εντολές μας προέρχονται από το παράρτημα 7 Οπότε αποφάσισα να δώσουμε κάποιες ε, διευκρινήσεις, ακριβώς επειδή υπήρξε και μια ανταλλαγή ε, ε, επιστολών με την εισηγήτρια και με την συνάδελφο Γιούτα Χάουκ, οπότε θα ήθελα ως πρόεδρος της Επιτροπής εδώ να πάρω θέση ως προς αυτό. Καταρχάς έχουμε την εισηγήτρια η οποία είναι ελεύθερη να δράσει ανεξάρτητα, ούτως ή άλλως πάντα έτσι το κάναμε και αυτό γίνεται και στις υπόλοιπες επιτροπές. Απ' την άλλη, η έκθεση δεν δεσμεύει μόνο ένα άτομο. Η έκθεση αυτή βεβαίως υπόκειται και, στις, στη βαρύτητα της, ε, των ομάδων του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, προφανώς ε, ζητά να ακολουθηθεί μια πολιτική διαδικασία έτσι ώστε ο εισηγητής, η εισηγήτρια, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, εν περιπτώσει, να μπορεί να επανασυνδεθεί με την ομάδα, με τους σκιώδεις εισηγητές και οι δράσεις που θα αναλυθούν να αναλυθούν με βάση την εντολή που υπάρχει. Οπότε προφανώς όλοι θέλουμε ο κάθε βουλευτής να μπορεί να ξεσκεί τα δικαιώματά του, αυτό δεν τίθεται καθόλου να αμφιβόλω. Βεβαίως όμως, ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ μπορώ να πω ότι εξ ονόματος της, ομάδας, της Επιτροπής ελέγχω του προπολογισμού μπορώ να πάρω το λόγο έτσι ώστε ακριβώς να ξανασυνδέσουμε λίγο την ομάδα με τους συντονιστές και με την εισηγήτρια. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού δεν μπορούμε να δράσουμε μεμονωμένα. Το δεύτερο πρόγραμμα ή το δεύτερη δράση που θα θέλαμε είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε ως ομάδα ή στα πλαίσια της συνολικότερης ε, ε, ε, βουλευτική, ε, ευρωβουλευτικής διαδικασίας ε, για να δούμε τι γίνεται με τους διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς όταν θέτουν θέματα ή ερωτήματα τα οποία δεν μπορεί να απαντήσει η εισηγήτρια του, της Επιτροπής Ελέγχου του Υπροπολογισμού. Δεν θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μα, προσπαθώ να είμαι λίγο προσεκτικός με την, ε, στη διατύπωσή μου. Απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βρούμε έναν δρόμο, μία λύση, έναν τρόπο να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία με αυτούς τους ευρωπαϊκούς φορείς. Οπότε ζητώ από όλους, ε, επιγόντως και βεβαίως και από την ε, εισηγήτρια Μακοβέη, να κάνει ό,τι μπορεί γιατί από αυτήν εξαρτάται, να έρθει σε επαφή με τους κοιόδης συγητές, έτσι ώστε στα πλαίσια αυτή τη κοινοβουλευτική διαδικασία να επιλέξουν μία ε, άγουσα που θα μα φέρει ε, πιο μπροστά αν τα καταφέρουμε αυτά και συνήθως ε, οι συγητές ε, μπορούν να συνοηθούν με τους ε, σκιώδες συγητές των άλλων ομάδων και καταφέρνουν να βρουν μια καλή συμβαστική λύση. Η εμπειρία λοιπόν στον οίκο μας δείχνει ότι οι συνάδελφοι που βρίσκονται πολλά, πολλές θητείες εδώ βοηθούν το Κοινοβούλιο γιατί στη συμφωνία βρίσκεται η δύναμή μας. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο με τις, ε, να είμαστε επικοδομητικοί και με τις ε, τροπολογίες και το Σεπτέμβριο να καταλήξουμε σε μια διαδικασία λήψης απόφασης, ψηφοφορίας που θα μας ε, οδηγήσει ένα βήμα παραπέρα. Ήθελα λοιπόν να τα πω αυτά γιατί Βλέπω ε, ότι δεν υπάρχει διάθεση τον επόμενο, τον Σεπτέμβρη ή τους επόμενους μήνες να τραβήξει κι άλλο αυτή η υπόθεση. Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εδώ στην ε, ομάδα μεταξύ μεμονωμένων ε, ατόμων. Δεν χρειάζεται να καταλήξουν στην ε, σύνοδο των ε, πρόεδρων, α πούμε, γιατί μόνο γιατί εκεί προφανώς θα δημιουργηθούν αρκετά έτσι, δυσίωνα σχόλια. Αυτό ήθελα να πω προς το παρόν στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να το διαχειριστούμε όλο αυτό το θέμα με μια τυπική διαδικασία και να την ολοκληρώσουμε θετικά. Δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Βλέπω εδώ με έναν κατάλογο ομιλητών. Η κυρία Μπροσμποά το θέλει το λόγο. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Γερμπράντι έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για μια πιο τεχνική ερώτηση προς την εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη. Μίλησε για ένα έγγραφο εργασίας ε, το οποίο εκπώνησε αλλά δεν είμαι πολύ βεβαίως για ποιο έγγραφο μιλάει. Οπότε, πριν μιλήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες, μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει για ποιο έγγραφο, μιλίας, για ποιο έγγραφο εργασίας μιλεί. Έχω έναν ε, μεγάλο κατάλογο μιλητών, έχουμε και την εισηγήτρια στον κατάλογο μιλητών, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Ε, ο κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την έκθεση της ε, συναδέλφου Μακοβέη, νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει καλά. Ε, το είδαμε και στην Επιτροπή, το έχουμε συζητήσει και στην Ολομέλεια. Ήταν αρκετά αντικρουόμενα τα αισθήματα, οι ψηφοφορίες. Ε, αυτό δεν είναι και ασύνηθες βέβαια όταν μιλούμε για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως η απαλλαγή και για τη δική μου την πολιτική ομάδα πρέπει να πω ότι ανησυχούμε για το πού τελικά θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί πέρα από την τυπική διαδικασία που έχει, οδηγεί, που εχει που ακολουθήσει η συγγήτρια, εμένα γενικώ με ανησυχεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία ε, για, αυτή, τις, για αυτούς τις υπηρεσίες τι θα κάνει. Ε, είχα και εγώ την απόψή μου, αλλά αυτό δεν είναι τώρα της παρούσης. Θα μπορούσε ίσως και η συγκίτρια να μας, πει αυτό, να μας το πει αυτό, αλλά η, ε, πώς μπορούν αυτοί, αυτές οι υπηρεσίες σε μια α, ε, ολομέλεια του Μαΐου, που μάλιστα τότε βγήκε η απόφαση, να α, παρεμβαίνουν τόσο σημαντικά και να έχουμε μία δεύτερη έκθεση το Σεπτέμβρη και λόγω ας πούμε των καλοκαιρινών διακοπών. Τελικά πόσο πολλοί μπορούν αυτές τις απαιτήσει που τους τίθενται να τις εκπληρώσουν. Κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι θετικό γιατί ε, θα γίνει ότι είναι ανθρωπίνος δυνατό, το οποίο βέβαια μετά θα τύχει και διαφόρων ερμηνεών για το αν όντω αρκούν οι προσεγγίσεις που έχουμε επιλέξει, οι προσπάθειες που έχουν, δίκη, ε, που έχουν γίνει. Η δική μου υπεποίθηση είναι ότι θα ληφθούν βεβαίως όλα αυτά υπόψη και θα δούμε αν όντω θα είναι τόσο θετικά τα πράγματα. Όλοι επιθυμούμε να είναι θετική εξέλιξη, αλλά δεν περιμέναμε ότι οι υπηρεσίες αυτές που γενικώ την χάνουν κριτικής που και που μέχρι στιγμής δεν, είχαν, δεν είχε συμφωνήσει το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, τι θα κάνουν για να μπορέσουν τελικά μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Οπότε δική μου, απέτηση, δική μου, δικό μου αίτημα μάλλον με βάση το ότι ακόμα σήμερα συζητούμε για το θέμα αυτό, για το πώς δηλαδή αυτά το, αυτό τον διοικητικό φόρτο, τον ε, ευρωπαϊκό, των ευρωπαϊκών υπηρεσιών μπορούμε να το μειώσουμε και όχι να τον αυξήσουμε, αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αυτό που κάνουν οι υπηρεσίες και αυτό που μπορούν να επιτύχουν πρέπει να το μετρήσουμε με βάση αυτό που αποφάσισε το Κοινοβούλιο, όχι πέρα από αυτό. Η εισηγήτρια ε, στέλνει συνέχεια ερωτήματα προς τις ε, υπηρεσίες. Ε, δεν είναι η δουλειά τους αυτή να απαντούν ερωτήσει, Η δουλειά τους είναι να κάνουν τη δουλειά τους ω υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών. Οπότε πραγματικά αναρωτιέμαι. για να είμαστε και δίκαιοι, μπορούν τελικά να εκπληρώσουν τις, τις υποχρεώσεις τους αυτές οι υπηρεσίες. Ή ξέρουμε όλοι ότι κάποιες από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει είναι αδύνατο να εκπληρωθούν. Θέλω να το πω αυτό ξεκάθαρα. Και θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ποιο είναι αυτό το διοικητικό άχθος που ε, επισύρει η, η θέληση του να επιτευχθεί αυτό που έχουν ως καθήκον αυτές οι υπηρεσίες και πόσο σημαντική είναι η δουλειά αυτών των υπαλλήλων που θέλουν να απαντήσουν και, τους, και ερωτήσεις των, ε, που τίθενται από τους ευρωβουλευτές γιατί θέλουν. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών υπεύθυνη και να εκπληρώσει την υποχρέωση που έχει για τον προπολογισμό που πρέπει να δοθεί σε αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να ελέγχει. Αλλά κύριε Πρόεδρε, το είπατε και εσείς, όταν κάτι είναι πολύ, είναι πολύ. Ας πούμε, η συγγήτρια ήδη κάνει προτάσεις για κάποια προγράμματα δράσης ε, των ε, υπηρεσιών και που πρέπει να τα αξιοποιήσουν, τότε πραγματικά αναρωτιέμαι ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Δεν θέλω να πω στην ουσία, απλώ στο γεγονός αυτό, από μόνο του αυτό λέει πολλά. Και με βάση το ότι Ίσως ε, να, υπάρχει και η παρέμβαση της συναδέλφου Χάουκ. Η ε, υπηρεσία ήταν ότι πρέπει να την αφήσουν να κάνει την ε, δουλειά της. Αυτή είναι η πρώτη τους δουλειά και η δεύτερη τους ας πούμε υποχρέωση είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής να, να επιβάλλουν ας πούμε, στο προσωπικό τους να απαντάει συνέχεια σε ερωτήματα ή να απαντάει σε καταλόγους που τους, αποστέλει ε, η, που τους αποστέλουν οι εισηγητές των διαφόρων ομάδων. Οπότε, οι συνάδελφοι που δεν είναι κάθε μέρα σε επαφή ε, με τις υπηρεσίες αυτές, καλό θα ήταν να το ψάξουν λίγο και να δούνε τι ακριβώς κάνουν αυτέ οι υπηρεσίε. Βεβαίω υπάρχει ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα, αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε κάποιου προσώπους αυτών των υπηρεσιών που θέλουν να απαντήσουν και θέλουν να παρουσιάσουν τη δική τους άποψη για το πώ δηλαδή τους επιβάλλουμε εμείς να, να ε, εκπληρώσουν τι τις υποχρεώσεις τους. Αυτά προς το παρόν, αλλά πραγματικά έχω ένα ερώτημα προς την κυρία Μακοβέη εσείς με την έκθεσή σας τι θέλετε να πετύχετε, ποιος είναι ο στόχος της έκθεσής σας. Έχω την εντύπωση ότι θέλετε στο τέλος αυτές οι υπηρεσίες να μην πάρουν την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Στάς έχει το λόγο. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τον κύριο Γκάιερ με πολύ προσοχή και σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ μαζί του. Είναι αλήθεια ασφαλώς ότι καθήκον μας είναι να θέτουμε πολλά ερωτήματα στις διάφορες αρχές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αρχές ε, τόσο σημαντικές ε, όπως η ασφάλεια των τροφίμων. Ε, γιατί όταν υπάρχουν, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε τέτοιου είδου ε, αρχέ, ε, μπορεί οι αποφάσει που θα λάβουν να είναι λανθασμένες. Πρέπει λοιπόν να θέτουμε τα ερωτήματα και να τι ενθαρρύνουμε να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Για ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν δεχτήκαμε την απαλλαγή για την αρχή των φαρμάκων και την αρχή της ασφάλειας των τροφίμων είναι η απουσία Έκθεση ε, ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο υπέβαλε τέτοιου είδους ε, έκθεση και για τις δύο αυτές αρχές και για την ΡΙΤΣ, τα χημικά, τις χημικές ουσίες και για την υπηρεσία ελέγχου της αεροπλοίας. Στις 29 Μαΐου του 2012, πιο συγκεκριμένα, υπέβαλε συστάσεις μέσω αυτών των εκθέσεων και ε, πιστεύω ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ελέγχου ε, του Προπολισμού θα έπρεπε να ζητήσετε την γνώμη του Ελληνικού Συνεδρίου και να κάνουμε γνωστή και τη δική μας γνώμη επί αυτών. Ε, γνωρίζω ότι ε, τα πορίσματα του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν, είναι, δεν, ε, δεν υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες και ενδεχομένως όχι όλες οι συστάσεις, αλλά με τη βοήθεια του Συμβουλίου και της Κομισιόν θα μπορούσαμε να τα αποκτήσουμε. Και θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά λοιπόν την γνώμη του Ελληνικού Συνεδρίου και το τι πιστεύει για το θέμα των τη σύγκρουση συμφερόντων σε αυτέ τι τέσσερι αρχέ και πιο συγκεκριμένα σε αυτέ τι δύο τι οποίε συζητούμε ε, σήμερα, ασφάλιση τροφίμων και φαρμάκων, για τι οποίε καθυστερήσαμε την απαλλαγή. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει ξεκάθαρα το πώς το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να οριστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τέτοιου είδου θέματα σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιου είδου ρυθμιστικό πλαίσιο ούτε για αυτέ τι ε, αρχέ ούτε και για πολλέ άλλε. Η κυρία Μακοβέη είπε ότι θα μπορούσαμε να βασιστούμε στι κατευθύνσει γραμμέ του ΩΣΑ, αλλά αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στι κατευθύνσει γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία των τρόπων εργασία για το μέλλον. Πρέπει να ε, μιλήσουμε με τον Διευθυντή και με το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό λόγο χρειάζεται ένα σχέδιο. Σχέδιο με διάφορες φάσεις. Συμφωνώ μαζί σου Γιάννης. Ε, δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά αν χάρη σε αυτή τη διαδικασία, την ε, συνομιλία, τις διαβουλεύσεις με τον Διευθυντή και με το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορούσαμε ε, να ετοιμάσουμε ένα προσχέδιο για την Ολομέλεια, τότε ε, αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει μέσω πρόθεσμα σε ένα πλαίσιο που θα βασίζεται σε συμφωνίες οι οποίες ε, θα έχουν συναυθεί στο πλαίσιο της ε, παραχώρησης της ε, απαλλαγής. Τόσο η αρχή των ευρωπαϊκών φαρμάκων όσο και η Ευρωπαϊκή Αρχή των Τροφίμων έχω την εντύπωση ότι έχουν καταλάβει το μήνυμα. Υπάρχει καλή θέληση και από τους διευθυντές τους και από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ασφαλώς υπάρχει και η αρχή του περιβάλλοντος, ε, η οποία είναι κάτι διαφορετικό, είναι διαφορετική περίπτωση. Το έχω πει και στην Ολομέλεια ότι αυτή η αρχή ε, περιβάλλοντος έχει κάνει πολλά λάθη. Και σοβαρά λάθη. Ε, θολές σχέσεις με μια μη κυβερνητική οργάνωση και άλλα προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να την, να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να ζητήσουμε ε, απαντήσεις και περιμένω ότι η, η μαζί με τους και ηγητές θα μας ε, βοηθήσουν να καταλάβουμε τι έχει γίνει ε, α, αλλά για τις δύο σημαντικές αρχές ε, αφενός και για την ε, αρχή περιβάλλοντος αφετέρου θα πρέπει ε, να μας υποβληθεί ένα πλαίσιο με συγκεκριμένες φάσεις και στάδια. Αυτό είναι το πολιτικό μας καθήκον. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Στάς. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αναφερθήκατε σε μένα ως πρόεδρο της Επιτροπής. Καταρχάς, η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχει ακόμα για το θέμα δηλαδή της σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν υπάρχει. Μας, το επέσ... την προσοχή ένα μέλος της Επιτροπής ότι δηλαδή ε, σχέδια αυτής της έκθεσης ε, του ελεκτικού συνεδρίου υπάρχουν οπότε εγώ στα περιθώριο της Ολομέλειας ήρθα σε επαφή με τον ε, πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου και του μίλησα για αυτό Εξ ονόματος της Επιτροπής ε, του ζήτησα το συντομότερο δυνατό να μας αποστείλει την επίσημη έκθεση. Οπότε νομίζω ότι η κριτική σας δεν έχει λόγο ύπαρξης γιατί έγινε αυτό που ζητάτε. Και επίσης ε, είπα να μας υποβάλουν την έκθεση. Εγώ δεν την έχω λάβει ακόμα την έκθεση αυτή του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνεδρίο δεν την έχει υποβάλει ακόμα. Επομένως το ερώτημα τώρα είναι τι, πώς διαχειριζόμαστε εκθέσεις που δεν έχουν υποβληθεί επισήμως. Πού στον ιστορικό κανονισμό υπάρχει η διάταξη που λέει πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες εκθέσεις τις οποίες ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου και κατά συνέπεια το ελεκτικό συνεδρίο δεν μας έχει υποβάλει. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο. Αν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα πολιτικό εργαλείο. Δεν γίνεται, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν μπορούμε εδώ μια επιτροπή να, να διαβουλεύεται επί μιας έκθεσης που δεν έχει επισήμως υποβληθεί. Υπάρχει και εσωτερικός κανονισμός και στο ελεκτικό συνέδριο και εκεί διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του. Το υποβάλλει την έκθεση όταν την υποβάλλει. Εμείς μπορούμε να το ζητήσουμε. Αν θέλετε μπορώ να το ξαναζητήσω εμεί δεν μπορούμε να ζητήσουμε να υποβληθεί η έκθεση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ο πρόεδρο Καλδέρα είπε ότι μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ θα υποβάλει αυτή την έκθεση. Αλλά δεν έχει και κανένα νόημα τώρα να κάνουμε ολόκληρα σενάρια για την έκθεση αυτή. Και τρίτον, τι θέλουμε τελικά να επιτύχουμε, όπω είπε και ο συνάδελφο Στάς. Οπότε προτείνω ε, επί τη βάση της έκθεσης ε, Μακοβέη και επί τη βάση της απόφαση ε, στην Ολομέλεια να ε, παρατείνουμε λίγο τη διαδικασία για τις υπηρεσίες αυτές, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι εδώ από την Επιτροπή ε, θεωρείται ότι είναι η τελευταία διαδικασία αυτή ε, απαλλαγής. Και αναρωτιέμαι, γιατί και στα επόμενα χρόνια θα έχουμε εκθέσεις για απαλλαγές και πάλι θα χρειαστεί να τις συζητήσουμε. Οπότε το ερώτημα είναι, επί τη βάση αυτών που έχουμε στα χέρια μας τώρα, τι κάνουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Αν τώρα τα δεδομένα λένε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή, τότε η Ολομέλεια μπορεί να πει δεν δίνεται η απαλλαγή. Αν πούμε ότι τα, αποτελέσματα, τα δεδομένα μας, ε, μας επιτρέπουν να δώσουμε την απαλλαγή, θα τη δώσουμε. Και μόλις δοθεί η απαλλαγή, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, θα δούμε πώς έχει η κατάσταση και το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα στην επόμενη διαδικασία απαλλαγής να ξαναυποβάλει τα επιχείρηματά του και να καταλήξει ίσως σε διαφορετική απόφαση. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτή η συζήτηση γιατί ε, έχει, ε, δημιουργείται με βάση μια εντύπωση ότι αυτό είναι το, το τέλος και δεν υπάρχει συνέχεια. Οπότε για τους συναδέλφους που θέλουν να ασκήσουν κριτική και σε μένα και στη γραμματεία παρακαλώ να την ε, αιτιολογήσετε αυτή την κριτική σας γιατί θέλω πραγματικά να ξέρω Ω πρόεδρο εγώ τι διαφορετικό θα έπρεπε να έχω κάνει. Γιατί απέναντι στο ελεγκτικό συνέδριο εγώ εκπροσωπώ τα συμφέροντά μα. Ζήτησα να μα υποβληθεί αυτή η έκθεση. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο και θέλουμε να παραμείνει ανεξάρτητο. Θα υποβάλει λοιπόν την έκθεσή του όταν την υποβάλει. Εμεί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαβουλευτούμε επί μια έκθεση που υπάρχει στα χέρια μα. Όχι επί μια έκθεση που βρίσκεται ακόμα στον εσωτερικό μηχανισμό του, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και ούτε θέλω να μιλούμε για σχέδια εκθέσεων ε, που ακόμα δεν είναι τελικά και για τα οποία έχει την, την ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ούτω ή άλλω, εμεί καλυπτόμεθα από τον ιστορικό μα κανονισμό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε την έκθεση. Μόλι μα έρθει η τελική έκθεση, θα τη συζητήσουμε. Αν δεν έρθει έγκαιρα για τούτη την ε, απαλλαγή, θα τη συζητήσουμε αργότερα. Ή μπορούμε να αρνηθούμε την απαλλαγή αλλά ούτως ή άλλως τη συζήτηση αυτή θα την κάνουμε πάλι για την επόμενη απαλλαγή. Οπότε παρακαλώ τον συνάδελφο Στάς να ε, αιτιολογήσει αν θέλει αυτές τις κατηγορίες που μας απίφθηνε. Το μόνο που θέλω είναι ε, η καλή συνεργασία με το, ε, με το ανεκτικό συνέδριο. Είχαμε πει, ξέραμε δεν θα είναι πριν το καλοκαίρι έτοιμη η έκθεση, αλλά ήδη είμαστε στο καλοκαίρι. Χρειάζεται, θα γίνει μια πρώτη συζήτηση το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, στο πλαίσιο μια καλή συνεργασία με το Ελληνικό Συνέδριο θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε ε, να επιταχύνουν λιγάκι. Ε, Όπω οι ποδηλάτε στο γύρο τη Γαλλία. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουν πιο γρήγορα πετάλι. Ε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Δεν σας επικρίνω, ούτε εσά ούτε την γραμματεία. Αυτό που ζητάω, ζητώ απλώς είναι ε, πολύ ευγενικά να ζητήσουμε από το Ελληνικό Συνέδριο να κάνει ό,τι μπορεί, να επιταχύνει λιγάκι. Ε, ε, έτσι ώστε το φθινόπωρο να είμαστε σε θέση να χορηγήσουμε αυτή την απαλλαγή. Ja, in aller Sachlichkeit, ich habe den Rechnungshof. Εξ ονόματος της, Επιτροπή, Επιτροπής μας, εγώ ζήτησα από το Ελεκτικό Συνέδριο να υποβάλει το συντομότερο δυνατό την έκθεση. Το, ο, ο πρόεδρος είπε ότι το νωρίτερο είναι μετά τις καλοκαιρινέ διακοπέ. Οπότε προτείνω μετά τις καλοκαιρινέ διακοπέ, να βάλουμε την έκθεση αυτή σε ένα ε, σημείο της ημερήσια διάταξη, να δούμε την έκθεση, να τη συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. το, η έκθεση αυτή δεν θα αφορά μόνο τρει υπηρεσίε, θα αφορά όλε τι υπηρεσίε. Οπότε ίσω να υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα και στοιχεία και θέματα που θα μπορούμε να συζητήσουμε στα πλαίσια της διαδικασία ε, απαλλαγή. Οπότε ίσω θα, θα βοηθούσε αυτό για να υπάρξει μια τελική άποψη στην Επιτροπή μα. Λοιπόν, έχουμε και άλλου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μιλητών. Θα ακούσουμε την κυρία Μακοβέη, μετά την κυρία Χέρτσοκ, την κυρία Βάιλερ, την Αγία Λασέντερ, Αντρέασεν και μετά ο κύριος Γκάιερ επίσης ζήτησε να, έρθουν, να μιλήσουν και οι παρόντες αν υπάρχουν εδώ από τις ε, υπηρεσίες αυτές. Ε, ξέρω ότι υπάρχει εκπρόσωπος μίας υπηρεσίας. Βεβαίως όποιος άλλος είναι εδώ και θέλει ευχαρίστως να πάρει το λόγο. Η κυρία Μακοβέη έχει πρώτα το λόγο. Παρακαλώ. Okay, Ίσως θα έπρεπε να απαντήσω καλύτερα στο τέλος, αλλά θα αρχίσω από τώρα να σας δίνω κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι η απόφασή μου να προτείνω αναβολή της απαλλαγής δεν ήταν πολιτικό ζήτημα. Πρόκειται για επαγγελματικό συμπέρασμα. Κάθε φορά λοιπόν που ακούω συναδέλφους να μιλούν για πολιτικά ζητήματα σε σχέση με τις συγκεκριμένε απαλλαγέ, εμένα προσωπικώ δεν μου λέει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό. Ε, αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα, κυρίω τη σύγκρουση συμφερόντων, τα οποία θέλουμε να επιλύσουμε προ όφελο των αρχών και των πολιτών. Κατόπιν. Αυτό είναι αυτό που έκανα αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ε, αρχίζουμε να συζητάμε ξανά τα πρώτη ε, ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έγινε, υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ανακοίνωσαν δύο μέρες ε, πριν από την ψηφοφορία ότι θα υπερψηφίσουν την απαλλαγή. Έχει καλώς. Αυτό το ξέρουμε. Ας συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα και είναι καθήκον μου να συνεργαστώ με τις υπηρεσίες. Δεν αρκεί απλώς να κάνουμε επικρίσεις στις εκθέσεις και να περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο να δούμε τι θα κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες και θα συνεχίσω με αυτό που αποκάλεσε ο κύριος ε, Στάς ε, χάρτες πορείας. Έχουμε αυτά τα έγγραφα εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκος και για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Να σας πω ότι κάθισα με το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πέντε ώρες και συζητούσαμε ε, αυτό το χάρτη πορείας και βλέπαμε τι υπάρχει, τι μπορεί να γίνει κλπ. Ήταν πολύ καλή η συζήτηση. Αντίστοιχα έγινε και με το Διευθυντή της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Και οι δύο λοιπόν αυτά αρχές, κατά την άποψή μου, θέλουν να αρχίσουν να εφαρμόζουν κάποια μέτρα προκειμένου ε, να μην υπάρχει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Δεν διαμαρτυρήθηκαν. Και γι' αυτό και εκπλήσωμαι για τα όσα ακούω αυτή τη στιγμή σήμερα. Δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία, συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Διαπιστώνω ότι κάποιοι συνάδελφοι διαμαρτύρονται όμως. Και όπως σας είπα, μίλησα και με τα διοικητικά συμβούλια ε, του κάθε οργανισμού και οι, τα διοικητικά συμβούλια με υποστήριξαν και δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε κάποιες από αυτές τις αλλαγές. Για να απαντήσω και στον κύριο Γκάγερ, παρά το γεγονός ότι μάλλον τη γνωρίζει την απάντηση, ε, προς τα που οδεύω, ε, εάν ε, δεν κάνω λάθο με ρωτήσατε να σας πω σαφέστατα ε, ε, ότι δεν θέλω να του δώσω την απαλλαγή. Όχι κύριε Γκάγερ, όπως σας είπα και στην προηγούμενη συνεδρία των συντονιστών και σε αρκετά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έστειλα ω συντονιστέ, ε, έχω επαναλάβει ότι θέλω να δώσω την απαλλαγή και θα ήθελα να πω και αυτό που είπα και στην αρχή με την προϋπόθεση ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου οι υπηρεσίες αυτές θα δείξουν ότι έχουν ξεκινήσει με αξιόπιστο τρόπο να εφαρμόζουν κάποια από τα μέτρα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο μέλλον και ότι δεσμεύονται να ακολουθήσουν αυτούς τους χάρτες πορείας. Αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν και πάλι, αυτή είναι η πρόθεσή μου. Και είμαι βέβαιη ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των ίδιων των υπηρεσιών και θα μπορέσουν να εργαστούν καλύτερα. Δεν ήθελα σήμερα να κάνω καμία μνήα στις επιστολές που έστειλαν οι άλλοι συνάδελφοι, διότι πραγματικά και πάλι επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να συζητήσουμε τι γίνεται τώρα με τις ίδιες τις υπηρεσίες ε, και πάλι να σας πω ότι αυτοί εργάζονται. Έχω την εντύπωση ότι οι ίδιοι είναι ικανοποιημένοι και να σας πω ότι ιδιαίτερα ο Οργανισμός Φαρμάκων ε, έχει δείξει ιδιαίτερη δέσμευση. Ο Διευθυντή. Ε, ξέφρασε την ίδια ακριβώ επιθυμία να κάνει αυτές τις αλλαγέ. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά από κοινού και να δοθεί απαλλαγή βάσει των προϋποθέσεων που σας ανέφερα τρεις φορές αν δεν κάνω λάθος. Αξιόπιστη εφαρμογή κάποιων από το μέτρο και δέσμευση να ακολουθήσουν αυτό το χάρτη πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επόμενος η κυρία Χέρτσοκ και μετά ο κύριος Γκερμπράντι και πάλι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω ογκρικά εφόσον μπορώ. Μιλούμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι είναι πραγματικά λυπηρό το ότι η συγκήτρια ανέβαλε την δουλειά που έπρεπε να γίνει με τους σκιώδες συγκητές και δούλεψε μόνο με τους συντονιστές. Πραγματικά αποκλείει τους σκιώδες συγκητές από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, η κυρία Μακοβέη είπε ότι το έγγραφο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια θέλει να το τροποποιήσει. Δεν θέλω να τη ρωτήσω, ε, θα μπορούσε να καταλήξει δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία τροποποίηση και σε ένα καινούριο έγγραφο, σε ένα καινούριο κείμενο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να καταλήξουμε σε μια έτσι αρμονία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και της εισηγήτριας σε ό,τι αφορά τις απόψεις μας. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό όταν ε, ε, όταν ζητούμε την συνεργασία με άλλες ε, ομάδες να την προσφέρουμε και εμείς ε, σε αυτές και να τη βελτιώσουμε. Η, η αρμόδια επιτροπή και οι υπόλοιπε επιτροπέ νομίζω ότι ήταν τερα... υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και στι υπόλοιπε επιτροπέ για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Και επίση ήθελα να ρωτήσω. Η Επιτροπή ΕΝΒΙ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υποβάλει μια γνωμοδότηση. Αν μπορεί, μήπως θα πρέπει να το κάνει πριν την ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Και ένα ακόμη ερώτημα έχω να θέσω σε ό,τι φορά τη διαφάνεια. Έχουμε μια ανταλλαγή επιστολών της εισηγήτριας με, συγκεκριμένες, ε, με μια συγκεκριμένη υπηρεσία, την οποία εμείς δεν έχουμε δει. Υπάρχει όμως αυτή η ανταλλαγή επιστολών. Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να δούμε αυτή την, αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή έθεσε η συγγήτρια ε, τα, ερωτήματα αυτά εξ ονόματος του Κοινοβουλίου ή τη Επιτροπής τη Κοκομπού στην υπηρεσία αυτή. Εμεί δεν έχουμε καθόλου καμία εικόνα. Δεν, είχαμε, δεν συμμετείχαμε στην όλη διαδικασία, δεν μπορέσαμε να θέσουμε τα ερωτήματά Μα δεν έχουμε καθόλου αίσθηση του πού βρίσκεται η κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να δούμε και η συγγήτρια εξ ονόματο τη ιδία ποιε ερωτήσει θέτει στι υπηρεσίε και επίση εξ ονόματο τη υπηρεσία ποιε ερωτήσει θέτει στι υπηρεσίε. Η Επιτροπή μας, σε σχέση με τα θέματα αυτά, δεν έχει καταλήξει ακόμα σε επίσημη θέση. Και ένα ερώτημα ακόμα. Έχουμε ψηφίσει τις αρχικές εκθέσεις. Σε αυτές είχαν τεθεί και τα ερωτήματα ε, υπάρχει δηλαδή αναλογικότητα ή δεν υπάρχει πια. Οι υπηρεσίες μας είπανε ότι έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, αλλά οι σκιώδεις συγητές ή οι συγγήτρια και οι συντονιστές μόνο μία ε, μέρα έχουν στη διάθεσή τους για να υποβάλουν τροπολογίες. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο, γιατί η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να τηρείται. Όλοι πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να μπορούν να κάνουν τις προτάσεις τους. Έχουν περάσει χιλιάδες ώρες για να καταλήξουμε τελικά σε αυτά τα, σε αυτά τα έγγραφα. Χιλιάδες ώρες δουλειάς. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Η εισηγήτρια Δύο μέρες μετά, ε, πριν την ε, συνεδρίαση μπορεί να μας ε, δίνει αυτά τα έγγραφα. Είναι σωστό αυτό σε εισαγωγικά. Μόνο δύο μέρες πριν η συγκίτρια έστειλε τελείω αυθαίρετα αυτά τα έγγραφα για το πόσες ώρες δαπάνησαν οι υπηρεσίε για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματά μας κτλ. Ε, Γενικώ δεν είναι απόλυτα σαφής η κατάσταση. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που μπορεί να θεωρούνται αρνητικές ή προσβλητικές για τις υπηρεσίες ε, πρέπει προφανώς να απομονωθούν. Ε, και έχω και ένα ερώτημα ακόμα, εξ ονόματος της σοσιαλιστικής ομάδας. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καθοριστούν κάποιοι κανόνες για το πότε υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όταν όμως αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν ακόμα ή επειδή δεν είναι σαφείς αυτοί οι κανόνες, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους θεωρήσουμε, ε, να τους ε, χρησιμοποιήσουμε αναδρομικά αυτούς τους κανόνες, γιατί αυτό ε, παραβιάζει την αρχή της ασφαλείας δικαίου. Η συγγήτρια έχει υποβάλει ένα κείμενο για την σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό το κείμενο είναι καλό. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό, γιατί επίσης τίθεται και το ερώτημα τι είναι τελικά πιο σημαντικό. Η λειτουργία αυτών των ε, υπηρεσιών ή αυτό που μας λέει η συγγήτρια και η δική της άποψη. Και επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω. Η συγγήτρια το σχολίασε ακροθυγός, ε, λέει, είπε κάτι για το πρόγραμμα δράσης ε, Υπάρχει κάτι που να είναι καινούριο, να υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο. Είναι, το σχέδιο δράση και ο δικό χάρτη που αναφερθήκατε είναι το ίδιο πράγμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χέρτσοκ. Ε, να συλλέξουμε λίγο τα ερωτήματα και μετά να ακούσουμε και την εισηγήτρια. Ο κύριο ε, Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ στη μητρική μου γλώσσα. Όταν φαντάζομαι την Επιτροπή μας, έχω κατά νου την προσοχή και τη φροντίδα, τη μέρημνα. Εμείς θέλουμε να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και αυτό ελέγχουμε. Μεριμνούμε ώστε να ε, τηρούνται κατά γράμμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να δρούμε κατά αυτόν τον τρόπο στις διαδικασίες που ακολουθούμε. Το Μάιο εγκρίθηκε η έκθεση στην Ολομέλεια. Και η απόφασή μας ήταν ότι ε, θέλαμε να δώσουμε την απαλλαγή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ε, έκθεση για την, ασφάλεια των για την υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων θέλαμε να υπάρξει η έκθεση και να παρακολουθήσουμε τα πράγματα για, να δούμε εάν το φθινόπωρο θα έχουμε ε, τη δυνατότητα να αλλάξουμε την απόφασή μας. Αυτή είναι η βάση συζήτησης. Και ε, με την ίδια αυτή προσοχή και ε, συνέπεια θα πρέπει οι υπηρεσίες να δεχτούν την απόφασή μας. Η απόφαση είναι ηλυμένη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία επί τη βάση της οποίας θα πρέπει να εργαστούν αυτές οι υπηρεσίες. Και τα ερωτήματα τα οποία τίθενται στο συγκεκριμένο ψήφισμα θα πρέπει να απαντηθούν. Και βάσει των απαντήσεων αυτών θα πρέπει να ε, ε, αποφασίσουμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο αν θα παραχωρήσουμε την απαλλαγή. Και εδώ θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση στην εισηγήτρια. Μου φαίνεται περίεργο το γεγονό ότι τίθενται ακόμα μια σειρά από ερωτήματα μετά από τι ερωτήσει οι οποίε ετέθησαν στο ψήφισμα του Μαΐου. Επί τη βάση ποιου πράγματο, ε, επί προσωπική ε, βάσεω, ε, θέσατε αυτά τα ερωτήματα, κυρία εισηγήτρια. Διότι ούτω ή άλλω το ψήφισμα είχε θέσει τα ερωτήματά του. Τι τελευταίε εβδομάδε λάβαμε και μια σειρά απαντήσει από τι υπηρεσίε. Και η γραμμή που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα μου το Μάιο θεωρώ ότι επιβεβαιώνεται στις απαντήσεις που λάβαμε. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν την άποψη της εισηγήτριας ε, στην ουσία για τις απαντήσεις που έλαβε μέχρι τούδε. Για, την, ε, τον οργανισμό φαρμάκων ε, πήρε μια πολύ καλή απάντηση, μας είπε, δεν άκουσα όμως την άποψή της για τις άλλες δύο υπηρεσίες. Βάσει λοιπόν του ψηφίσματος του Μαΐου, αυτές οι τρεις υπηρεσίες μας απάντησαν. Ε, τι άποψη έχει η συγγήτρια για αυτό. Από εκεί και πέρα. Ο χάρτης πορείας, ο οποίος αναφέρθηκε από την εισηγήτρια. Ε, να σας πω ότι εκπλήσουμε λίγο. και πάλι έχει να κάνει με το πόσο διεξοδικοί είμαστε. Επί ποιες βάσεως ε, ετοιμάσατε αυτό το νοδικό χάρτη. Ε, είναι η προσωπική σας άποψη. Το κάνετε εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, το κάνετε εξ ονόματος της ε, Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικώς δεν συμμετείχα ποτέ σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας, στην οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε χάρτης πορείας και σας δώσαμε εντολή ως εισηγήτρια να εκπονήσετε αυτό το χάρτη πορείας. Σε ποιο βαθμό λοιπόν έχετε μεριμνήσει ως προς αυτό. Τρίτον, ε, η ζημία που προκαλείται στη φήμη αυτών των υπηρεσιών. Πρόκειται για δύο για τρεις συγγνώμη, ισχυρές υπηρεσίες, τους έχουμε χωρίσει σημαντικά καθήκοντα, Πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες ε, ε, διεξάγουν σημαντικά καθήκοντα, αλλιώ δεν θα υπήρχαν, ε, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξη. Και ε, ο λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση είναι ακριβώ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτοί οι οργανισμοί. Είναι λοιπόν προ το συμφέρον μα να έχουν εξαιρετική φήμη αυτέ οι υπηρεσίε, όχι μόνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι επικρίσεις δεν είναι η άποψη της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, αλλά είναι προσωπικές απόψεις της ίδιας της εισηγήτριας, οι οποίες είναι εις βάρος κάποιων υπηρεσιών. Και είναι σχεδόν αδύνατο να αναστρέψουμε την κατάσταση. Για το ψήφισμα που εγκρίθηκε το Μάιο, σκεφτείτε εάν ε, ήταν το ψήφισμα αυτό το οποίο προκάλεσε τη ζημία και δυσφήμισε ουσιαστικά τις υπηρεσίες αυτές ή είναι οι προσωπικές σας απόψεις σας. Ε, από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο αυτή την έκθεση για τη σύγκρουση συμφερόντων. Και εγώ προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Ε, συμφωνώ και με τις παρατηρήσεις της δικές σας κύριε Πρόεδρε, ότι η, έκθεση υπάρχει όταν γίνεται επίσημη δημοσίευσή της. Επομένως δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε κάποιος να δει εκ των προτέρων αυτή την έκθεση. Στους διαδρόμους ακούγεται ότι κάποιοι ε, προβουλευτές διαθέτουν την έκθεση και κάποιοι όλοι όχι. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Ε, μπορούμε παρόλα αυτά να πιέσουμε το ελεγκτικό συνέδριο ώστε να ζητήσουμε να ετοιμάσουν την έκθεσή του στο συντομότερο δυνατόν. Το ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι το έχετε ζητήσει, ίσως θα μπορούσατε να επαναλάβετε το έτοιμά σας. Η Επιτροπή μας μαζί με τον υπεύθυνο από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, ε, λήξει η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για τη διαδικασία της απαλλαγή, θα μπορούσε ίσως να κάνει μία συνεδρίαση και να συζητήσει την έκθεση αυτή. εγώ ξεκινάω βέβαια από την προϋπόθεση ότι τον Ιούλιο ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε λάβει αυτή την έκθεση. Ίσως και στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και να μπορέσουμε να συνεδριάσουμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε την έκθεση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύγκρουση συμφερόντων και ε, δεν θεωρώ ότι μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία απαλλαγής εάν δεν έχουμε διαβάσει την έκθεση και δεν έχουμε συζητήσει το περιεχόμενό της με το ελεγκτικό συνέδριο. Περιμένω λοιπόν την απάντησή σας κύριε Πρόεδρε. Να σας απαντήσω άμεσα. αν έχουμε την έκθεση εγκαίρω, θα την ε, συζητήσουμε και θα δούμε αν όντω μπορούμε να οργανώσουμε μια ειδική συνεδρίαση ή όχι. Αλλά βεβαίω αυτό πρέπει να το δούμε και με την προθεσμία που έχουμε για τι ε, τροπολογίε, την 6η Σεπτέμβρη. Θα δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Μέχρι στιγμή λοιπόν δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα έχουμε την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, οπότε αυτά μπορώ να σα πω. Η κυρία Γκρέσλε μετά η κυρία Σεν και μετά η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε λιγάκι να αφήσουμε την σκόνη να κατακάτσει. Η συνάδελφος Μακοβέ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ε, διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό το διαπιστώσαμε ήδη δύο φορές. Το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων στις υπηρεσίες ε, και πέρσι Ασχοληθήκαμε ακριβώς με το ίδιο πράγμα. Και τα προηγούμενα χρόνια πάλι ασχοληθήκαμε με το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα της ΣΥΠΟΛ. Πάντα λοιπόν υπάρχει μια υπηρεσία για την οποία οι προσεγγίσεις που υπάρχουν είναι διαφορετικές. Σημαντικό τώρα είναι να μην κάνουμε κάτι που θα μας αποδυναμώσει. Η συνάδελφος Μακοβέη είναι η συγγήτρια για το Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι για την εξέβρεση λύσεων που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου ήταν η παράταση. Εγώ προσωπικά με την απαλλαγή για την, για την υπηρεσία ασφάλειας τρομίμων και, την... και των φαρμάκων θα μπορούσα να τη δεχτώ. Οι άλλες δύο τώρα υπηρεσίες έχουν πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε και δεν προσπαθεί να το λύσει και η συγκήτρια. Το θέμα μας είναι όμως να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα του, της, της σύγκρουσης συμφερόντων με έναν ευρωπαϊκό τρόπο. Οι ειδικέ επιτροπές πρέπει να δούνε πραγματικά το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων, να αφοσιωθούν σε αυτό. Αυτή η διαδικασία είναι μακροσκελής. Πρέπει να ζυγίσουμε τι θέλουμε. Προφανώ θέλουμε να υπάρχει βιομηχανική γνώση σε αυτέ τι υπηρεσίε. Αλλά αυτέ οι υπηρεσίε μάλλον το, θα πρέπει να είναι τόσο σαφές το πλαίσιο με στο οποίο θα λειτουργούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε καν η μικρότερη δυνατή αφιβολία ότι μπορεί να υπάρξει επιρροή από κάποιον εξωτερικό. Και ακριβώς επειδή είναι ε, θέμα υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορούμε να αφήνουμε να πλανώνται ε, αμφιβολίες για τη δουλειά που κάνουν αυτές οι υπηρεσίες. Θέλουμε λοιπόν σαφείς διαδικασίες και θέλουμε και σαφείς διατάξεις. Αν δούμε τώρα τι έχουν κάνει και πώς έχουν προχωρήσει οι υπηρεσίες, Υπάρχει, ούτως ή άλλως οι εμπειρογνώμονες τους δίνουν την δήλωση συμφερόντων ας πούμε, οι οποίες όμως δεν εξετάζονται ποτέ. Ε, δεν υπάρχει κανένας που να εξετάζει ε, εις βάθους αν θα μπορούσε να υπάρχει έστω και μια αμφιβολία σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω λοιπόν ότι η κυρία Μακοβέη λέει ακριβώς αυτό που αποτελεί το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε να, να μην το συζητήσουμε. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα τέλο πάντων τελεσίδικα δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά είμαι αντίθετη να, να μην δώσουμε την απαλλαγή στι υπηρεσίε επειδή έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Προφανώ έχουν το πρόβλημα αυτό. Και η ε, υπηρεσία για τα φάρμακα και η, για, τα, για τι χημικέ ουσίε έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά όσο δεν μπορούμε να λύσουμε εμεί το πρόβλημα, δεν μπορούμε να του αρνου, αρνούμαστε την απαλλαγή. Οπότε πραγματικά το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ε, σε βάθος. Ξέρω ότι πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα όλα αυτά. Ξέρουμε ότι ζητούμε από τις, ε, πολλή δουλειά από τις υπηρεσίες γιατί τους, τους στέλνουμε προφανώς ε, πολλές ερωτήσεις. Είναι καλό που τους στέλνουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις γιατί είμαστε και εμείς σοβαροί πολιτικοί αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια σωστή λύση. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Οπότε ζητώ και ξαναζητώ να συνεργαστούμε. Έτσι κάνουμε, έτσι κάναμε πάντα για να προχωρήσουμε σε αυτή την έκθεση. Εγώ προσωπικά ως συντονίστρια ε, έθεσα πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι η κυρία Μακοβέη ε, διέθεσε τόσο γρήγορα τις, ε, τις δικές της προτροπολογίες για την έκθεσή της. Αν μπορούσε ο καθένας από εμά να συνεργαστεί για να κάνουμε κάποιες τροπολογίες, να δούμε ποιες θα είναι αυτές που θα υποβληθούν, να δούμε αν μπορούμε να τις δεχτούμε ή τι άλλο μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνω τον θυμό, καταλαβαίνω την ενόχληση όλων, γιατί ο καθένας από εμά πάντα βρίσκει ως αντίπαλο αυτό ακριβώς το, το πρόβλημα. Υπάρχει όμως το πρόβλημα. Και είναι ακριβώς τόσο έγκαιρα ε, έχουν υποβληθεί αυτές οι τροπολογίες της κυρίας Μακοβέη, οπότε μπορείτε όλοι να δείτε αν θέλετε να τις δεχτείτε, αν μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί της ή αν θέλετε να υποβάλλετε εσείς οι ίδιοι ε, τροπολογίες. Η κυρία Ανδρέας αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την Επιτροπή και θα το επαναλάβω. Η απαλλαγή αφορά το παρελθόν. Έτσι χορηγείται. Όχι το μέλλον. Και οι φορολογούμενοι θέλουν να γνωρίζουν μας ζητούν να εγκρίνουμε τη διαχείριση των δικών τους χρημάτων στο παρελθόν, αλλά όχι στο μέλλον. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς ως Επιτροπή έχουμε παγιδευτεί από μόνοι μας. Δηλαδή, ε, σκάψαμε το λάκκο μας εν στο παρελθόν. Ε, έχουμε αναβάλει για άλλες υπηρεσίες, για άλλους οργανισμούς την απαλλαγή. και επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης. Όμως η κατάσταση στο μέλλον θα βελτιωθεί, όχι στο παρελθόν. Οπότε αυτή η αντιφατική ε, τάση να ε, θέλουμε με το παρελθόν να λύσουμε τα προβλήματα του μέλλοντος ε, δεν έχει νόημα γιατί ούτως ή άλλως μόνο υποσχέσεις και σχέδια δράσης έχουμε για το μέλλον. Έχουμε παγιδευτεί λοιπόν σήμερα σε αυτή την κατάσταση και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αμηχανία όταν μιλάμε για την αξιοπιστία των οργανισμών. Έχουμε ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και στο παρελθόν. Πέρσι το ίδιο κάναμε με την ε, ΣΥΠΟΛ. Αναβάλαμε την απαλλαγή και δώσαμε την απαλλαγή 6-8 ε, μήνες αργότερα επί τη βάση πάλι υποσχέσεων για το μέλλον, ε, για το ε, πώς θα πήγαιναν τα πράγματα στο μέλλον στο συγκεκριμένο οργανισμό και όχι σε σχέση με τις ανεπάρκειες και αποτυχίες του παρελθόντος. η έγκριση της διαχείρισης γίνεται σε σχέση με την απόδοση στο παρελθόν, όχι στο μέλλον. Αν συνεχίσουμε ε, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα ε, τύχουμε ποτέ του σεβασμού των φορολογουμένων. Ε, γελοί θα γίνουμε και γελιότεροι θα είμαστε όταν υπάρχουν συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο που μπορούν να γράφουν στις συγκεκριμένε υπηρεσίες και να τους λέμε ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε ερωτήματα. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να σκεφτούμε λιγάκι το πώς συμπεριφερόμαστε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Γιάννα Sí, eh, ε, Συνήθως δεν συμφωνώ με την κυρία Ανδρέα Σένα, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε πολλά από όσα είπε. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διάκριση ανάμεσα ε, στη, στα, τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, της επιτροπή Προπολογισμών και, και τις ε, ε, Αποκεντρωμένη Είναι μια κατανομή που δημιουργεί τέτοιου είδου συγκρούσει. Ε, όμως ο δημοσιονομικό έλεγχο έχει ω στόχο να ελέγξει ε, ακριβώς την υλοποίηση του, ε, την εκτέλεση του προπολογισμού. Το, η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το εντοπίσουμε, αλλά δεν είναι δικό μας καθήκον να το επιλύσουμε. Υπάρχουν ε, άλλες ε, επιτροπές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τώρα, να επιστρέψω στη δική μας διαδικασία. έγινε μια ψηφορία το Μάιο. Σήμερα σύμφωνα με τα όσα εξήγησε η κυρία Μακοβέη, ε, έχουν γίνει πλέον μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, τροπής, τρόπου λειτουργίας κλπ. Οπότε ε, έχουμε μια έκθεση, ε, μια δεύτερη έκθεση. Δεν είναι δυνατόν η δεύτερη έκθεση να είναι η ίδια με την πρώτη. Πρέπει να υποστηρίξω την κυρία Μακοβέη. Θα έπρεπε να ήμασταν πιο σοβαρή και να έχουμε υποβάλει μια καινούρια πρόταση που να συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις βελτιώσεις. Διότι τι θα πούν οι πολίτες όταν δουν να επαναλαμβάνει την ιστορία, η ίδια ιστορία. Ενώ οι ίδιοι μέσω ίντερνετ ενδεχομένως θα μπορούσαν να διαπιστώσουν ότι έχουν ήδη γίνει αλλαγές, έχουν γίνει βελτιώσεις. Οι πολίτες αν διαβάζουν τη δική μας έκθεση όμως θα νομίζουν ότι δεν συνέβη τίποτα και θα γελάνε μαζί μας. Αναγνωρίζω επίσης τον ε, πειρασμό ε, από επικοινωνική πλευράς του να θίξουμε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Ε, το έχουμε δει επανειλημμένως και σε πολύ ανώτερες θέσεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα με έναν επίτροπο. Το ζήτημα όμως είναι ότι εμείς δεν μπορούμε ε, να βάλουμε στον ίδιο σάκο όλες τις ε, αρχές, όλους τους οργανισμούς ε, και να θίξουμε τη φήμη τους. Η υπηρεσία του περιβάλλοντος είναι αυτή που έχει τα περισσότερα προβλήματα. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Έχουμε δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν και συνεχίζουμε. Το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι το, το διαχειριστικό του σχέδιο είναι εξαιρετικό και αν πλέον έχουμε κάποια προβλήματα που πρέπει να λύσουμε με την Επιτροπή, δεν είναι δυνατόν αυτά να τα φορτώσουμε και σε όλες τις υπόλοιπες ε, ε, αρχές. Ε, οι εκθέσεις των αρχών αυτών είναι δημόσιες, συγκρίνονται, διαβάζονται. Ίσως υπάρχει ένα θέμα σύγκρουση συμφερόντων, εντάξει μπορεί, για ένα άτομο, αλλά δεν είναι ένα μόνο το άτομο το οποίο κάνει αυτές τις εκθέσεις που συντάσσει, συντάσσει Ε, τέλος να πω ότι ε, θέλω να κάνω έκκληση προς τον κύριο Γκέιερ. Ε, θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα. Δεν είναι δυνατόν ε, να ε, δεσμεύουμε 10 μήνες από το χρόνο ενός υπαλλήλου ε, για να απαντήσει στα ερωτήματά μας σε σχέση με τη σύγκρουση φερόντων ενός ανθρώπου. Ε, είναι δυσανάλογα μεγάλος ο χρόνος ε, που σπαταλάτε, η ε, πόρη, το δυναμικό που σπαταλάτε για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου δεν είναι τόσο σημαντικό. Θα έπρεπε να διαθέτουμε δυνατότητες άλλες σύγκρισης και επιβεβαίωσης. Αυτή η δυσαναλογία με ενοχλεί θα πρέπει να είμαστε ικανοί να ε, καθορίσουμε κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και ταυτόχρονα κανόνες για την ε, τήρηση της αναλογίας. Να μην είναι δυσανάλογο πολύ ο χρόνος, πολύ ο χρόνος που σπαταλάτε για τέτοιου είδους ζητήματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Χέρτσοκ και μετά να ακούσουμε τους εκπροσώπους των ε, υπηρεσιών εφόσον το επιθυμούν. Η κυρία Χέρτσοκ έχει και πάλι το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάθε ε, βουλευτής έχει το δικαίωμα να, στέλει, να θέτει ερωτήματα. Αλλά όταν τα θέτει εξ ονόματος της Επιτροπής, προφανώς χρειάζεται και την υποστήριξη της Επιτροπής. Και αυτή τη φορά δεν υπήρχε η στήριξη της Επιτροπής. Ε, συμφωνώ με την συνάδελφο, θα, ε, ούτως ή άλλως πρέπει να τηρήσουμε την αναλογικότητα, την ε, τάξη, αλλά εδώ δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις, σαφείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κρεμάσουμε κάποιον χωρίς να έχουμε λόγο που τον κρεμάμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς κανόνες. Γι' αυτό έχω άλλο ένα ερώτημα. Είναι σημαντικό να δούμε η άποψη της ΑΦΚΟ ποια είναι. Μια που βρισκόμαστε στα πλαίσια της συναπόφασης. Θα ήταν νομίζω σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χέρτσοκ. Ερώτημα τώρα προς τους εκπροσώπους των υπηρεσιών. Ε, η κυρία, η καθηγήτρια Μακλέιντ είναι εδώ. Παρακαλώ, να σας δώσω το λόγο. Ε, ή, εν πάση περιπτώσει, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ανδρέας Πόρτ, εκπροσωπώ την ε, υπηρεσία φαρμάκων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουμε κι εμείς. Δύο λόγια ήθελα μόνο να πω για την υπηρεσία ε, φαρμάκων, γιατί προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλων υπηρεσιών, ε, γιατί είναι διαφορετικές από τη δική μας. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό για μένα να διαπιστώσω ότι με την, ε, έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με την εισηγήτρια και αυτό δεν έγινε μόνο ε, λόγω της εισηγήτρια, αλλά και λόγω της συνεργασίας που έχουμε και με την Επιτροπή σας και με το Κοινοβούλιο που πάντα είναι, ε, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντούμε όλα τα ερωτήματα και να εφαρμόζουμε οτιδήποτε μέτρο χρειάζεται. Με την υπηρεσία φαρμάκων είχαμε την τύχη και πέρσι να λάβουμε με αναβολή βέβαια την, ε, την απαλλαγή μας. Οπότε έχουμε μάθει αρκετά από το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Αλλά εδώ δεν μιλούμε μόνο για σύγκρουση συμφερόντων, κυρίες και κύριοι. Μπορεί αυτό όντως να είναι το πιο σημαντικό θέμα. Αλλά αν δείτε την έκθεση που υπάρχει από τον Μάιο και που υπάρχει και σήμερα εδώ, περιλαμβάνει, ε, σε αντίθεση με άλλα χρόνια, πολύ περισσότερα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την διαδικασία που, με την οποία κινείται η υπηρεσία μας και αυτή χρειάστηκε να αλλάξει. Αυτό σημαίνει μεγάλο άφθο για τις υπηρεσίες μας. Όλα τα μέτρα που είχαμε λάβει μέχρι στιγμή στην υπηρεσία έφταναν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να Α πούμε, για να απαντήσουμε σε μια επιστολή ενό βουλευτή, όχι τη συζητητέ, ενό βουλευτή, έπρεπε να κάνουμε διάφορε αναλύσει, διάφορε έρευνε για να απαντήσουμε μόνο σε, ένα, σε μια επιστολή. Αυτό κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ για να σα δώσω μια τάξη μεγέθου. Ποια μέτρα δηλαδή είναι αυτά που είχαμε, που πάρει. Ε, Επίση, πολύ σημαντικό είναι, σε σχέση με το θέμα αυτό, ότι χρειάζεται ε, μία αξιόπιστη ε, διαδικασία μέτρησης για το, ε, σε εισαγωγικά μέτρησης για το τι απαιτεί και από μας το κοινοβούλιο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε η κυρία Αντρέασεν, μπορούμε να μάθουμε από το παρελθόν και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μαθήματα για το μέλλον, ώστε να έχουμε αξιόπιστα μέτρα. Και επίση σημαντικό είναι για τις ε, υπηρεσίε τα μέτρα για τα οποία σας ενημερώνουμε και τα οποία έχουμε λάβει να είναι γνωστά και στο Κοινοβούλιο και να λαμβάνονται υπόψη. Έχουμε πάντα την εντύπωση ότι ε, πάντα θέλετε να υποβάλλετε νέες εκθέσεις για νέα μέτρα. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Είναι σημαντικό να ε, βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο ως ε, ε, πολιτικό παίκτη και να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές του, αλλά από την άλλη πρέπει να μην υπονομεύεται και η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη που έχετε εμείς, εσείς σε εμά και εμείς σε εσά. Και επίσης να πω κάτι άλλο για το ελεγκτικό συνέδριο και τη σχετική έκθεση που συζητήθηκε με αρκετή ένταση. Η υπηρεσία φαρμάκων είναι, βρίσκεται σε διαδικασία αμφισβήτηση τη έκθεση του ε, ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Από τον Ιούνιο ήταν έτοιμη η ε, ε, έκθεση αυτή. συζητούν τέσσερι υπηρεσίε την έκθεση αυτή με, την, με το ελεγκτικό συνέδριο και από όσο ξέρουμε στην τελική, του μορφή, στην τελική της μορφή η έκθεση αυτή θα υποβληθεί μέσα ή προ το τέλο του Αυγούστου. Ευχαριστώ κύριε Πόρτ. Έχει κανένας άλλος να πει κάτι από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ προέρχομαι από τον Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Οργανισμό. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να πάρουμε και εμεί το λόγο. Μερικά πράγματα θα ήθελα να πω και εγώ. Δεν εμφανιστήκαμε για τόσο ε, πολύ στη συζήτηση, αλλά προφανώς ε, έχουμε κάποιο πρόβλημα στα μάτια της συγγήτριας. Ε, χάρηκα που έγραψε στις 27 Ιουνίου η κυρία Μακοβέη, ευχαριστώντα ε, ευχαριστώντας και αναγνωρίζοντας την ε, συνεργασία μας και υπό το φως αυτής της ε, ανταπόκρισής μας και των ερωτήσεων στις 10, 19 Απριλίου, στις 13 Μαΐου και στις 13 Ιουνίου προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας για ε, την, το σύγκρουση συμφερόντων και για το πρασίνισμα γνωρίζετε ότι υπήρξαν πάρα πολλές φορές ε, ε, αποστολές, 126, ε, για να δουν κατά πόσο ισχύουν αυτά που ισχυριζόμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Γκρέσλε και την κυρία Αντρέα Σεν ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και μιλούμε για την απαλλαγή στο παρελθόν, που αφορά το παρελθόν δεν έχουμε σχέδιο δράσης, ούτε χάρτη πορείας, αλλά υπήρξαν κάποιες δράσεις, πέντε που μας αφορούσαν, διαδικασίες για τη σύγκρουση συμφερόντων, κανόνες αποδοχής, ε, ε, του διευθυντή και τη σχέση του με άλλους ε, οργανισμούς, ε, Όσον αφορά τώρα την πολιτική κατάρτιση. Ε, ζητώ συγγνώμη, Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις και ήμουν διαθέσιμη ευχαρίστως να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις. Αλλά δυστυχώς αυτό που δεν μπορώ να κάνω δεν μπορώ να απαντώ σε κατηγορίες ε, από τον τύπο ε, με ερωτήσεις που μοιάζουν με τις δικές Κάνω ό,τι μπορώ να ε, συνεχίσει η λειτουργία του οργανισμού μας. Προσπαθήσω, προσπαθώ να αυξάνω την αυτοπεποίθηση του προσωπικού μου και προσπαθώ να είμαι ο καλός πολίτης, για να το πω έτσι. Για παράδειγμα, στο ψήφισμα της 10ης Μαΐου ε, ζητείται περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη ε, σχέση με ε, το κοινό εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε μας προς αυτό. Εμείς δεν προσπαθήκαμε ποτέ να αποκλίνουμε από τους οικονομικούς κανόνες. Ευχαρίστως να απαντήσω ερωτήσεις σχετικά. Κάναμε ό,τι μας συζητήσατε. Οπότε θα ήθελα να πω ότι αν κρινόμαστε για το παρελθόν, Ρωτήθηκε για παράδειγμα το Διοικητικό Συμβούλιο αν ε, ενημερώθηκε. Ναι, βεβαίω ε, ρωτήθηκε. Αν θέλετε τώρα ε, να επικρίνετε αλλά να επικρίνετε τα θέματα τη σύγκρουσης για τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων, είπαμε ότι ο Οργανισμό θα κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά του επιστήμονε. πάλι λέει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ενθαρρύνει, να, ενθαρρύνει την συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να υπάρχουν συνεργασίε και για να να συμμετέχουν όλο και περισσότερο οι πολίτες. Ε, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ζητού συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω εκ μέρου ε, του προσωπικού μου. Ε, προσπαθούμε πάρα πολύ να λάβουμε αυτή την απαλλαγή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά, συγγνώμη, ε, έχω συγκινηθεί πολύ. Ε, δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο συγκινημένη, ίσως γιατί βλέπω, ξέρω ότι βγαίνουμε και στο διαδίκτυο, αλλά 1.400 ώρες δαπανίσαμε να απαντούμε στα ερωτήματά σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το παρελθόν. Ε, θα προσπαθήσω για το μέλλον. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω και περισσότερες απαντήσεις. Και συγγνώμη πάρα πολύ που ε, συγκινήθηκα και αναστατώθηκα τόσο. Äh, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακλέιτ. Το πιο σημαντικό είναι στην Επιτροπή εδώ να θυμόμαστε ποιος είναι ο στόχος της όλης διαδικασίας ε, απαλλαγής και ότι πρέπει να μείνουμε στα πλαίσια μιας πολύ αυστηρής εντολής. Να δω αν είναι κανένας άλλος εκπρόσωπος εδώ της ΕΦΣΑ ή κάποιες άλλες υπηρεσίες για να σας δώσουμε το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Thank you, Mr. Uh, ε, ονομάζομαι Αλμπέρτο Σπανιόλη. Ε, είμαι επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλισης των Τροφίμων. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω κατά κάποιο τρόπο τα σχόλια των συναδελφών των δύο προηγούμενων αρχών υπηρεσιών που μίλησαν. Η ΕΦΣΑ επίσης συνεργάστηκε πλήρως, προσπάθησε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κατόπιν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν των επακόλουθων ε, ερωτήσεων της συζητήτρια. Ε, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μέχρι το τέλος. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά για μας απέτησαν σημαντική αφιέρωση πόρων, ε, επένδυση σε πόρους και σε χρόνο. Παρ' όλα χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα λύνει τα προβλήματα, ιδιαίτερα το θέμα του σύγκρουση καρόντου, γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε αυτή την επένδυση. Αναγνωρίζουμε ότι η απόφαση της Επιτροπής σας στο τέλος της διαδικασίας θα βασίζεται σε τρία βασικά, σε τρία βασικά τύπους εγγράφων. Πρώτον, το, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που την περιμένουμε όλοι. Δεύτερον, το νοδικό χάρτη, το πρόγραμμα εργασίας ή πρόγραμμα δράσης όπως και να το πούμε και σε αυτό συνεργαζόμαστε και τρίτον οι απαντήσεις που έχουμε ήδη δώσει στην έκθεση και στις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την 10η Μαΐου. Θέλουμε να μας ε, καθισχάσετε κατά κάποιο τρόπο ότι όλη αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει ε, θα ληφθεί υπόψη. Γιατί καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι ε, συντάσσουμε πολλά έγγραφα, μεγάλο όγκο σελίδων και δεν εξετάζονται λεπτομερώς. Για παράδειγμα, μέσα σε αυτά τα έγγραφα έχουμε ήδη δώσει εξηγήσει, λεπτομέρειε εξηγήσει για τα νέα μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει του τελευταίους μήνες σύμφωνα με τη νέα πολιτική ανεξαρτησίας και τους νέους εφαρμοστικούς κανόνες, τους οποίους εφαρμόζουμε τώρα πλέον. Με βάση αυτούς τους κανόνες ε, ε, κάναμε ε, τον έλεγχο των νέων εμπειρογνωμόνων. δεχτήκαμε πολλές κριτικές τα περασμένα χρόνια για τις παλιές μας διαδικασίες. Ε, ακούστηκαν διάφορα, διάφορες διαδόσεις, ε, ισχυρισμοί και απαντήσαμε σε όλα αυτά. Ελπίζω όλες μας αυτές οι απαντήσεις να ε, μελετηθούν λεπτομερώς και σοβαρά και να ληφθούν υπόψη στις τελικές σας αποφάσεις. Τούτου λεχθέντος, να δώσουμε και άλλες απαντήσεις αν χρειάζεται. Πάντως, οι ήδη απαντήσεις που έχουμε δώσει είναι αρκετές. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μια λύση που θα είναι αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τις παρεμβάσεις των υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Χάουγκ. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, δεν ήθελα να πω τίποτα, αλλά η κυρία Μακλάιντ ε, έτσι όπως παρενέβη και με όλα αυτά που έχει ζήσει και όλα αυτά που μας είπε με παρακίνησε να πάρω και εγώ το λόγο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος, ε, ε πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ελέγχων. ήμουνα υπεύθυνη εισηγήτρια για όλες τις υπηρεσίες. Και τώρα βεβαίω, η, ε, την εργασία τη η ε, διαθεσμική ομάδα. Ε, ήμουν πρόεδρος της διαθεσμικής ομάδας για τι υπηρεσίε. Κατά την άποψή μου νομίζω ότι κάναμε αρκετά επιτυχή δουλειά. Βεβαίως... Ε, ακόμα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λύσει και η Κομισιόν αλλά και ε, εμείς οι ίδιοι πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Τώρα, γιατί πήρα το λόγο. Γιατί η κυρία Μακοβέη προφανώς ε, δεν το έγραψε βέβαια στην έκθεση, αλλά προφανώς προσπάθησε στον τύπο να μιλήσει με μισές αλήθειες, με ενδείξεις, με κάποιες προσωπικές προσβολές και με επιθέσεις να κάνει πολιτική. Και αυτό εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο μπορώ να σας το, να σας το πω. Ε, το ότι κάποιο θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του και θέλει να κάνει τη δουλειά του με αφοσίωση και με ζήλο, δεν μπορεί να αντιδρά με τέτοιο συναισθηματισμό και να θεωρεί ας πούμε ότι όταν κάποιος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και προσπαθεί να απαντήσει σε ψευδή ε, σχόλια προφανώς είναι λογικό να έχει έτσι τόσο πολλές ε, ε, τόσο συναισθηματικές εξάρσεις. Ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, λέει η κυρία Γκρέσλα, γιατί δαιμονοποιείται η συνάδελφος. Θα ήθελα να πω το εξή. Αυτές οι αντιδράσεις ε, δεν είναι σωστές. Εδώ ή θα συζητήσουμε μεταξύ μας και οι διευθυντές των ε, υπηρεσιών γι' αυτό είναι κλεγμένοι για να συζητούν ή θα αφήσουμε τη συζήτηση. τέτοιου είδους Αντιδράσει, ε, προφανώ αλλάζουν λίγο την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμω, θα ήθελα να πω το εξή. Αυτά που υπάρχουν στο τραπέζι εδώ και για την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την οποία με την οποία ασχολήθηκα εγώ ε, έχουμε το θέμα των ε, ταξιδιών στην Καραϊβική, της χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι θέματα σοβαρά τα οποία θα καλυφθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Πραγματικά λοιπόν θέλω να, να ζητήσω μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Γιούτα, καλό θα ήταν να πάρουμε κι εμείς αυτές τις πληροφορίες που έχεις, αλλά παρακολούθησα λίγο εγώ αυτές τις πληροφορίες που μας ανέφερες και θα ήθελα πραγματικά το πρόβλημα αυτό να μην, να μην το μετατρέπουμε σε, ένα, ε, σε μια κατηγορία απλώς των συναδέλφων μας. Ε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να λύσουμε το πρόβλημα ιδιαίτερα με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει τα ερωτήματα που υπάρχουν να απαντηθούν και να μείνουμε εκεί. Τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Η κυρία Μακοβέη και πάλι έχει το λόγο. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ. πολύ συναισθηματισμός και ομολογώ ότι εγώ δεν έχω συναισθηματισμούς. Εμένω στα επαγγελματικά εδώ. Έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να σας πω εν συντομία δύο-τρία πράγματα και να απαντήσω στα όσα ακούστηκαν. Η σύγκρουση των συμφερόντων είναι στη δικαιοδοσία της Επιτροπής μας. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των πόρων, τη διαχείριση των κονδυλίων, και έχει σχέση και με τα πλήρη αποτελέσματα και τις δραστηριότητες ε, των οργανισμών αυτών. Κατόπιν, μέτρα για την πρόληψη ή τη διαχείριση της σύγκρουσης των συμφερόντων είναι τα συνήθι μέτρα που λαμβάνουμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι αυτά που συζητήσαμε και με τον Οργανισμό Φαρμάκων και με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Αν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στη βιομηχανία και γίνονται και πυρογνώμονες ε, στους οργανισμούς, τότε θα πρέπει να είναι γνωστό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ε, εργάζονται στην τάδε εταιρεία, συμμετέχουν στην τάδε ομάδα του οργανισμού και γνωμοδοτούν για το χ προϊόν ή για το χ έχει Επομένως, η διαφάνεια και αντίστοιχα στοιχεία είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε είναι ε, η πάγια πρακτική μας εδώ και χρόνια σε αυτούς τους οργανισμούς ε, που ε, εξειδικεύονται και σε θέματα αυτά και μας ενδιαφέρει η σύγχρονη η σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτή είναι και η εντολή μας. Ε, έχουμε και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που περιμένουμε να έρθει εδώ στην Επιτροπή μας και να μας πει ε, τι φρονεί το ελεγκτικό, συνεδρίο, ε, το ελεγκτικό συνέδριο για τη σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, όσον αφορά τη φήμη των οργανισμών, Κύριε Γκελμπράντε, στόχο μου είναι να βελτιώσω τη φήμη των οργανισμών, διότι υπάρχουν πολλοί ισχυρισμοί στα μέσα μαζική ενημέρωση και από συγκεκριμένου μη κυβερνητικού ε, οργανώσει προ ε, και τον Οργανισμό Φαρμάκων και κυρίω τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Προφήμων και θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω τη φήμη αυτών των οργανισμών, βοηθώντα του να λύσουν τα προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων. Αν δείτε τι. Ε, πάμπολες αναφορές που υπάρχουν κυρίως για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Προφήμων και θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, και θα δείτε ότι πριν από κάποιες μέρες ε, η επικεφαλής ε, της, ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων συμμετείχε σε κάποιο γνωστό λόμπι και υποχρεώθηκε να παραιτηθεί μία μέρα πριν δημοσιοποιηθεί. Στόχος μου λοιπόν είναι να βοηθήσω τους οργανισμούς αυτούς να βελτιώσουν το πρόβλημα, να λύσουν το πρόβλημα και να βελτιώσουν τη φήμη τους. Ε, και με τα χαράς ε, να πάω να τους βοηθήσω, να σταθώ στο πλάι των ε, επικεφαλής των οργανισμών, να μιλήσω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να σας πω τι καταφέραμε στο τέλος. Η απαλλαγή, είπατε, αναφέρεται στο παρελθόν. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν θέλουμε μόνο να αναλάβουμε δεσμεύσεις για το μέλλον. Θέλουμε να υπάρχει εφαρμογή, να υπάρχει τουλάχιστον μία αξιόπιστη απόδειξη ότι έχουν ξεκινήσει αυτά τα μέτρα. Και από τα όσα έχω λάβει εγώ στοιχεία και από τον Οργανισμό Φαρμάκων και από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εγώ έχω τέτοιε ενδείξει. Και να σα πω ε, ότι ναι και οι γραπτέ σα απαντήσει και όλα τα στοιχεία που μα δίνετε προ τον κύριο τη ΕΦΣΑ ε, θα ληφθούν υπόψη και θα γίνουν οι κατάλληλε τροπολογίε. Η έκκληση που κάνω προς όλους είναι να μην αποθαρρύνουμε τους οργανισμούς να συνεχίσουν αυτό το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει. Και δύο λόγια τώρα για τα όσα είπε η κυρία Χάουγκ. Για τους ισχυρισμούς αυτούς. Εγώ στην αρχή της συζήτηση δεν αναφέρθηκα στην επιστολή που αποστήλατε εσείς προς τους οργανισμούς, αλλά με υποχρεώνετε να το κάνω τώρα. Στείλατε επιστολή προς τους τρεις οργανισμούς χωρίς να διαβουλευτείτε ποτέ με την εισηγήτρια και τους είπατε ότι κάποια πράγματα υπερβαίνουν την εντολή μου. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η στάση βεβαίως, αλλά εγώ δεν ήρθα να σας ρωτήσω γιατί το κάνατε. Ο καθένας από μας έχει το δικό του τρόπο εργασίας και πραγματικά δεν περιμένω και απάντηση, διότι δεν σκοπεύω να σας απαντήσω κι εγώ τίποτα. Κάντε ό,τι νομίζετε. Θέλετε να στέλνετε επιστολές, στείλτε. Και μια τελευταία παρατήρηση για τον οργανισμό περιβάλλοντος. Όπως σας είπα, μίλησα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχω απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρόκειται για σοβαρά προβλήματα και θα ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει αμέσως μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να προληφθεί η σύγκρουση συμφερόντων, κάποια μέτρα που αφορούν και την ε, αποδοχή του εκτελεστικού διευθυντή οποιασδήποτε άλλης θέσης σε άλλους οργανισμούς, ε, έλεγχος ε, μεταφορών κονδυλίων μεταξύ γραμμών προϋπολογισμού και ούτω καθεξής. Ναι, βεβαίως έχουν ληφθεί μέτρα και εξετάζοντας και το επίπεδο εφαρμογής ε, τον Αύγουστο, όλα αυτά θα αντικατοπτρίζονται και στις τροπολογίες. Αλλά για όλους αυτούς τους συναισθηματισμούς, εγώ θα ήθελα να μην είμαστε συναισθηματικοί και να πούμε δύο πράγματα για τις ασυνέπειες που υπάρχουν στην αλληλογραφία μας με τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Τρία παραδείγματα θα σας δώσω και σας διαβεβαιώ όλους ότι έχω γραπτά στοιχεία για όλα όσα θα σας πω. Όταν ρώτησα αν υπήρχε κάποια μη κυβερνητική οργάνωση επιτόπου που στεγάζεται στα γραφεία του οργανισμού, μου απάντησαν όχι. Και όταν διαπίστωσα ότι στην ιστοσελίδα μιας συγκεκριμένης μη κυβερνητική οργάνωση η διεύθυνσή τους είναι ίδια με του Οργανισμού περιβάλλοντος, έλαβα μέτρα ώστε να απομακρυνθούν. Πρόκειται για δημόσιο έγγραφο και στην, ε, στα εγγένεια του συγκεκριμέ, συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που στεγάζεται στα γραφεία του Οργανισμού Περιβάλλοντος ήσασταν εκεί και δώσατε μια αναρκτήρια ομιλία. Γνωρίζετε λοιπόν ότι στεγάζονται στα κτίριό σα. Άλλο παράδειγμα. Μας γράψατε Κυρία Μακοβέη. Δεν είμαστε δικαστήριο, κυρία Μακοβέη. And we this, we we know... Και θα μείνουμε απλώς στη διαδικασία απαλλαγή. Σας παρακαλώ λοιπόν, ε, κυρία Μακοβέη να τηρήσετε και το χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώστε την παρέμβασή σας και μετά θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Θα σας στείλω όλα αυτά τα έγγραμμα ξανά, παρά το γεγονός ότι τα έχω ξαναστείλει πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, αλλά θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Όταν ε, ο διευθυντής ε, έγινε μέλος του Συμβουλίου του Earth World, Είχαμε στοιχεία, είχαμε στοιχεία για τον Νοέμβριο και μετά στην ιστοσελίδα είδαμε ότι ε, εντάχθηκε στο Earth World το 2009. Μετά από μία ώρα βέβαια άλλαξαν τα στοιχεία στην ιστοσελίδα. Απλώς σας λέω ότι όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα. Υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις και εγώ θέλω να έχω μία τίμια σχέση με άλλους. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο με τον Οργανισμό Φαρμάκων και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Θέλω να συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τους τρεις οργανισμούς, καλή την πίστη, να λάβω υπόψη όλα τα αποτελέσματα και τις δεσμεύσει τους μέχρι τα μέσα Αυγούστου και για άλλη μια φορά, συνάδελφοι, θα σα στείλω όλα αυτά τα έγγραφα και τις ε, τροπολογίες μου πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσπάθησα να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, που σημαίνει ότι μπλέχτηκε τελείως τώρα το χρονοδιάγραμμά μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν σημαντικό να συζητήσουμε εντελεχώς το θέμα αυτό, γιατί προφανώς θα χώναμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σημαντικό είναι σε αυτή τη συζήτηση να παραμείνουμε στον έλεγχο του προπολογισμού και στην απαλλαγή και για το κατά πόσο μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια που δίνει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό. Μην ξεχνούμε ότι όλοι είμαστε σε ε, θεσμικά ε, όργανα. Παρ' όλα αυτά, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πάντα άνθρωποι και πρέπει να τους ε, μεταχειριζόμαστε με την απαραίτητη διπλωματία και ανθρωπιά. Ε, οπότε ε, η ανθρωπιά είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην την ξεχνάμε. Ας την έχουμε πάντα υπόψη μας σε όλους τους πολιτικούς μας αγώνες. Ας μην μιλούμε μόνο για νούμερα. Προφανώς πρέπει να κάνει ο καθένας τη δουλειά του, αλλά Γι' αυτό προσπαθήσαμε, να, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σήμερα εδώ, αλλά ήθελα απλώ να πω ότι δεν έχει, δεν έχει κανένα νόημα σε μια διαδικασία απαλλαγή να μπαίνουμε σε τόσο μεμονωμένα στοιχεία για τα οποία ούτως ή άλλως είναι πολύ περιορισμένος και ο χρόνος και δεν μπορούμε και να δημιουργήσουμε ένα σαφές πλαίσιο. Η κυρία Μακλέιντ μας είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν 1.400 ώρες εργασίας για να απαντηθούν οι ε, ερωτήσεις των βουλευτών. Είναι δικαίωμα των βουλευτών, των βουλευτών να, δίνουν, να θέτουν ερωτήματα. Αλλά προφανώς ε, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας και το τι σημαίνει να απαντηθούν αυτά τα ε, ερωτήματα. Έχουμε λοιπόν τώρα μία πρόταση διαδικασίας. Εάν το επιθυμείτε, θα κάνουμε άλλη μία έξτρα ε, συνεδρίαση για, τις, ε, για τους οργανισμούς. Θα βρεθώ εγώ με τους συντονιστές, αν θέλετε θα έρθω σε επαφή μαζί τους μετά τις ε, ε, καλοκαιρινές διακοπές, να έρθουμε εδώ και δύο μέρες ας πούμε να ασχοληθούμε μόνο με τους οργανισμούς. Σήμερα δεν έχουμε επαρκή χρόνο. Ε, είχαμε ε, προετοιμαστεί μόνο για 45 λεπτά συζήτησης, χρειάστηκε τελικά πολύ περισσότερη ώρα, οπότε προφανώ. Έχουμε και τον ε, ε, κύριο Στόιμπερ ε, καλεσμένο, οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με το χρονοδιάγραμμά μας. Έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, για τις εκθέσεις της απαλλαγή. Ας μείνουμε στην διαδικασία μας. Η κυρία Μακοβέη είπε ότι θα έρθει σε επαφή με τους σκιώδης ηγητές και θα συνεργαστεί μαζί τους. Το είπε σήμερα. Το, το υπογραμμίζω, κυρία Μακοβέ, υπογραμμίζω αυτό που είπατε. Είσαστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με τους σκιώδει συγκητέ. Η ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου. Οπότε μπορούμε αυτό το σημείο προς το παρόν να το κλείσουμε. Προς το παρόν. Κλείνουμε το σημείο αυτό δεν ξέρω, θέλει κάποιο άλλο το λόγο, γιατί αλλιώς μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να συνεχίσουμε παρακάτω. Η κυρία Χέρτσοκ θέλει το λόγο, κάτι διαδικαστικό. Πρόεδρε, ένα σχόλιο. Δεν πήραμε απάντηση για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ερώτημα θέσαμε. Ούτε εγώ, ούτε η σκιώδη οι υπόλοιποι. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι ε, λογικό αυτό να δημιουργείται τέτοιο χάος και κάποια στιγμή κάπου η κυρία Μακοβέη θα μας δώσει κάποια απάντηση. Ε, συγγνώμη, αυτό δεν είναι δυνατό να συμβαίνει. Για, διαδικαστικό, για τον εσωτερικό κανονισμό, τι, ε, κυρία Γκρέσλε, όχι, ο κύριος ε, Σάρβαμα έχει το λόγο. I will be very, very brief. Θα είμαι σύντομος. Πρώτον, συμφωνώ πλήρως με τα όσα είπε ο πρόεδρος. Δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Αλλά, δεύτερον, εξίσου σημαντικό, δεν θα καταλήξουμε κάπου πριν αποκτήσουμε μια ενιαία ερμηνεία του κατά πόσον η σύγκρουση φερόντων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Αν ερμηνεύουμε διαφορετικά ή δίνουμε διαφορετική απάντηση σε αυτό το θέμα, τότε θα κάνουμε κύκλους. Αυτό είναι μια παρατήρηση. Δεν προτείνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά το λέω αυτό ως νέο μέλλον. Θα είμαι σκιός ηγητής του ΕΛΚ για τις ε, αρχές για την επόμενη χρονιά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το κατά πόσον η σύγκρουση, το, συμφερόντων εμπίπτει στην εντολή και στα καθήκοντα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε, να κλείσουμε το θέμα αυτό. Είπαμε ότι κάποιοι σκιώδεις ηγητές θα έρθουν σε επαφή με την εισηγήτρια. Σημειώνουμε ότι κάποια ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Η ε, εισηγήτρια περιμένει τις απαντήσεις από, το, από τις υπηρεσίες. Ε, προφανώς και οι σκιώδεις περιμένουν την εισηγήτρια να τους δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Θέλετε όλα αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε στην Επιτροπή ή να πούμε ότι η εισηγήτρια πήρε το λόγο και συζητήσαμε τα θέματα αυτά όσο πιο εις βάθος μπορούσαμε και ότι τώρα μπορούμε να συμφωνήσουμε όπως είχαμε, συμφωνήσει, όπως είχαμε προβλέψει, να υποβληθούν δηλαδή τροπολογίες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου και μετά να συνεχίσουμε με τη γνωστή δημοκρατική διαδικασία και να το λύσουμε. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Νομίζω ότι Συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν έτσι και κλείνουμε το σημείο αυτό μετά από μια πραγματικά πολύ ζωντανή συζήτηση. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους ε, προέδρους, ε, τους εκπροσώπους των ε, Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Τώρα, προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Η Επιτροπή Θέλετε να, να φέρουμε το σημείο με τον κύριο Στόιμπερ λίγο πιο μπροστά στην ημερήσια διάταξη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε άρα τώρα τον κύριο Στόιμπερ και μετά θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Εντάξει. Ωραία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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, Συνάδελφοι, να σας πω ότι αμέσως μετά την παρουσίαση του κυρίου Στόιμπερ θα κάνουμε την ε, ψηφοφορία, δηλαδή γύρω στις 5. Ο κύριος Στόιμπερ έχει ένα μισάωράκι για να μας αφιερώσει. Οπότε ε, έχουμε λίγο καθυστερήσει με την ε, μερίσια διάταξή μας. Τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά στις πολιτικές συζητήσεις. Συζητήσαμε λοιπόν πώς ε, μπορούμε να έτσι, ποινικοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες. Ε, ο κύριος Στόιμπερ θα, θα μας μιλήσει για το κόστος της γραφειοκρατίας, για, την, για το βάρος που έχει αυτό στους Ευρωπαίους φορολογουμένους. ο διοικητικός φόρτος είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Σύμφωνα με το παράρτημα 7 είμαστε υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα των δαπανών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βεβαίω, ε, στην ομάδα εργασία σα έχετε υποβάλει πάρα πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει για το πώ αυτή η επιβάρυνση των ε, Ευρωπαίων φορολογουμένων μπορεί να μειωθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Γι' αυτό χαίρομαι που μπορούσαμε να σας φέρουμε σήμερα ε, ε, εδώ να μας μιλήσετε για τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν πώς μπορεί κανείς να φρενάρει τη γραφειοκρατία. Νομίζω το χρειαζόμαστε επιγόντως αυτό και ίσως ε, θα μπορούσαμε, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πολλές φορές, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δούμε το θέμα της, της επίδρασης του ευρωπαϊκού προπολογισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μεν, αλλά να δούμε και την επιπτώση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και στου Ευρωπαίου φορολογούμενου και πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό χωρί όμω να επιβαρύνουμε με νέα διοικητικό άχθο ε, τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ, Δόκτωρ Στόιμπερ, σήμερα. Χαίρομαι που είσαστε ενώπιον της Επιτροπής ε, Ελέγχων του Προπολογισμού και μπορείτε να μας ε, παρουσιάσετε την άποψή σας παρακαλώ το, χρησιμοποιήστε καλύτερα το αριστερό σας μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Μάλιστα, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, το φθινόπωρο του 2008 ήρθα πρώτη φορά στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να κάνω μια παρουσίαση ε, επίσημη ε, για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κάνουμε και εμεί ό,τι μπορούμε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά δεν είχα την εντύπωση ότι το 2012 θα ξανάρθω για να κάνω την ίδια παρουσίαση. Η Κομισιόν βεβαίω. Από το 2010 στο 2012 παρέτεινε την, την εντολή μου, οπότε θα υπάρξει μάλλον κι άλλη παράταση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί πραγματικά πάρα πολύ αυτό το θέμα της γραφειοκρατίας και της απάλληψής της να το διαχειριστεί πολύ σοβαρά. Στην παρούσα κρίση, κύριε Τόερερ το είπατε, η μείωση της γραφειοκρατίας μπορεί να, να συμβάλλει σημαντικά στην περισσότερη ανάπτυξη και στην απασχόληση. Γιατί ακριβώς Σημαίνει αυτό οικονομική ανάπτυξη, οικονομικά προγράμματα χωρίς ιδιαίτερο κόστος, γιατί μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη περίπου 1,5%. Έχει προτείνει και η Κομισιόν αρκετά πράγματα, αν όλα αυτά λοιπόν μπορέσουν να εφαρμοστούν και ευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς. Βεβαίως το θέμα του ε, ευρώ στις 29 Ιουνίου συζητήθηκε και εκεί συζητήθηκε ακριβώς η, ε, η, η σημασία που έχει η μείωση της γραφειοκρατίας και βεβαίως ε, και εγώ ως ε, πρόεδρος της ε, Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου έκανα μια πολύ σοβαρή ανταλλαγή απόψεων με τους προσώπους των εθνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή είτε στη Ρώμη, είτε στο Βερολίνο, είτε σε άλλες χώρες πρέπει και αυτοί, οι αρχές δηλαδή, να συζητήσουν και μεταξύ τους για το τι κάνουν οι ίδιες οι αρχές για να εφαρμόσουν την οδηγία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει επαρκώς. Ε, και πρέπει να πω επίση ότι η μείωση τη γραφειοκρατία ε, και για άλλου λόγου είναι ιδιαίτερο υπαρξιακό ζήτημα, γιατί πολλέ μικρέ επιχειρήσει λόγω ακριβώς όλων αυτών των διατάξεων αισθάνονται πνιγμένες και οι εμπειρογνώμονε που πήραν μέρο και οι εμπλεκόμενοι φορεί που ήρθαν στην ομάδα ε, είπαν τι απόψει του. Και είναι πραγματικά τρομακτικό ότι μία σειρά επιχειρήσεων ε, και μάλιστα στην ε, Ευρώπη έχουμε μείωση, έχουμε έλλειψη μάλλον αυτοαπασχολούμενων ατόμων βλέπουν όλοι αυτοί ότι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες η γραφειοκρατία αυξάνεται. Είναι, υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά παραδείγματα τα οποία και εγώ από μόνο μου παρόλο που ήμουνα ε, στην, ε, στο ιστορικό της Γερμανίας ενεργό σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή δεν τα, δεν τα γνώριζα τόσο καλά. Και υπάρχει και άλλη μία τρίτη διάσταση τη ε, μείωσης της γραφειοκρατίας. αφήσουμε, αφήσουμε το θέμα του ευρώ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως αυτό είναι θέμα που, έχει, που ξυπνάει πολύ τα αίματα. Αλλά όλοι εσείς όπως και εγώ ξέρουμε ότι και στις χώρες και στην Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Πενελούξ υπάρχει ένα ερώτημα. Όταν ρωτάει κανείς τους πολίτες τι συνδέεις με την ε, Ευρώπη, τι σημαίνει η Ευρώπη για σένα, 40% των πολιτών λένε «Ε, ένα τέρας μακρινό, ε, χωρίς καθόλου φιλικό προς τους πολίτες, που παίρνει μόνο αποφάσεις με αυτό ακριβώ, με αυτή την απάντηση πρέπει να, την, πρέπει να, την, να ασχοληθούμε, πρέπει να τη δούμε σοβαρά. Αν δηλαδή 40% των πολιτών θεωρούν ότι αυτό είναι η Ευρώπη και όχι αυτό που πραγματικά είναι η Ευρώπη, τότε νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Περίπου 20% στο σύνολο της, ε, των Ευρωπαίων ε, πολιτών ε, έχει διαφορετική άποψη ας πούμε, μεταξύ Πορτογαλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας κτλ. Δηλαδή η άποψη τους, της γραφειοκρατίας είναι διαφορετική για κάθε χώρο. Οι Πορτογάλοι δεν βλέπουν ότι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, οι Βρετανοί το βλέπουν διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ένα πέμπτο των πολιτών της Ευρώπης όταν τους ρωτάνε τι σημαίνει για σένα Ευρώπη λένε γραφειοκρατία, ένα τέρας γραφειοκρατίας κτλ. Αυτό είναι πρόβλημα για μας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το βάρος της ε, ε, εφαρμογής των ευρωπαϊκών ε, κανόνων και διατάξεων είναι στην πρώτη θέση. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θεωρούν ότι επιβαρύνονται. Και βεβαίως αυτό σημαίνει επιβάρυνση για 23 εκατομμύρια ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη που σημαίνει επιβάρυνση 100 ε, δις ευρώ. Η Κομισιόν έλαβε μια απόφαση στα τέλη του 2007 και έλεγε ότι μέχρι το τέλος του 2012 θα είχε μειώσει τη γραφειοκρατία κατά 25%. Και αυτό λέει ότι θα μπορέσει να σπρώξει και την ανάπτυξη. Δηλαδή θα υπήρχαμε ανάπτυξη περίπου 1,5% στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή θα είχαμε εξοικονόμηση 150 δις ευρώ. Εμείς, η ομάδα υψηλού επίπεδου, από το 2008 κάναμε πάνω από 300 ε, προτάσεις στην Κομισιόν με δυναμικό εξοικονόμησης περίπου 140 δις ευρώ. Από αυτά 30 δις ευρώ Δηλαδή, ε, ε, καταφέραμε να ε, ωφελήσουμε τις, επι, τις ε, επιχειρήσεις κατά 30 δις ευρώ μέσω των αποφάσεων Κομισιών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Οπότε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να ε, διευκολύνουμε τις ε, επιχειρήσεις. Ε, γιατί κάποιες φορές οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ληφθούν και αυτό δυσκολεύει τις επιχειρήσεις. Δηλαδή η αλλαγή των αποφάσεων στην Ευρώπη διαρκεί 7 χρόνια κατά όρο και αυτό είναι πάρα πολύ μακρά περίοδος. Για μένα είναι πάρα πολύ μακρά και πρέπει όντως να προσπαθήσουμε αυτά τα 7 ε, χρόνια να τα, να τα μειώσουμε. Και πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχουν ε, ε, βεβαίως προτάσεις που πάνε προς την τελείως λάθος κατεύθυνση. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις όντως είναι δύσκολο γιατί το πεδίο έντασης μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να σπάσει. Η γραφειοκρατία για μένα ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη ένταση. Ε, δηλαδή ε, εσύ είσαι υπέρ της ε, ευθύνης του κάθε ατόμου, της, του κινδύνου που θέλει να, να αναλάβει ή είσαι υπέρ, είσαι υπέρ του να υπάρχει ασφάλεια μέσω των νόμων, δηλαδή μέσω διοίκησης, άρα γραφειοκρατία. Ασφάλεια λοιπόν απέναντι στην ελευθερία είναι πάντα μια εξίσωση που ε, δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει και η βεβαίως η ψηφιακή ε, διάσταση και πρέπει να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Τώρα, για την ασφάλεια των ε, ταξιδιωτών, για την ασφάλεια των μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει τους, τις περιόδους ξεκούρασης. Ο οδηγός δηλαδή κάθε εβδομάδα δεν μπορεί να οδηγά πάνω από 56 ώρες. Δηλαδή κάθε μέρα όχι παραπάνω από 9 ώρες. Και 4,5 ώρες πρέπει να κάνει, κάθε 4,5 ώρες πρέπει να κάνει διάλειμμα. Αυτό τα έχουμε ορίσει μέσω του ε, ψηφιακού ταχογράφου. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε ότι τηρούνται αυτοί οι κανόνε, στα διάφορα ταξίδια με ε, φορτηγά πάνω από 3,5 τόνου πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό ταχογράφο. Το κόστος είναι περίπου 4.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως θέλει να υπάρξει ε, ασφάλεια. Απαιτεί λοιπόν ε, από οποιονδήποτε μικρό, μικρομεσαίο οδηγό, μεταφορέα κτλ. που μπορεί ας πούμε μια φορά ή δύο φορές το μήνα να χρησιμοποιεί το φορτηγό του και να κάνει ας πούμε 50, 60, 80 χιλιόμετρα για να παραδώσει κάτι, ακόμα και αυτός πρέπει να έχει ηλεκτρονικό ταχογράφο. Και μάλιστα οι άνθρωποι λένε είσαστε τρελοί, δεν, δεν γίνονται αυτά. Για, τους, για, τον, για, τους, για να εξυπηρετήσουμε τους λόγους της ασφάλειας τους επιβαρύνουμε ακόμα, ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι, αυτές είναι τυπικές περιπτώσεις, τυπικά παραδείγματα που μας έχουν πει οι άνθρωποι που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Και πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της, ε, της ψηλού επίπεδου έχει κάνει πρόταση ήδη από το 2008. Το 2009 μαζί με την εφημερίδα Bild και την Sun είχαμε κάνει μάλιστα ε, ένα διαγωνισμό για το ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον project για τη μείωση του, ε, της γραφειοκρατίας. και ο ηλεκτρονικό ταχογράφο είπα, ε, είπαν ε, όσοι απέντησαν ότι ε, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν κάποιο ταξιδεύει πάνω από 150 χιλιόμετρα. Για μικρέ δηλαδή και μικρομεσαίε επιχειρήσει, Μόνο όταν η, ε, τα ταξίδια είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα χρειάζεται ο, ηλεκτρονικό, ταχογράφο, Μίλησα με τον Ταγιάννη, μίλησα με τον Κάλλα, με τον Ταγιάννη, μάλιστα σχεδόν συμφωνήσαμε. Μετά αυτό έφυγε, ήρθε ο Κάλλα. είπε ξανά θα τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή και καταλαβαίνετε ότι αυτή, αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Και τώρα τελικά καταφέραμε να υπάρξει μια λύση όπου η Κομισιόν λέει εντάξει όχι 150 χιλιόμετρα αλλά για όλους όσους κάνουν ταξίδια πάνω από 100 χιλιόμετρα θα, ε, ε, θα χρειάζονται ταχογράφο. Που σημαίνει ότι αντί για 50 ή 100 χιλιόμετρα, ε, ναι, δεν θα έχουμε ε, όριο ανά ε, χιλιόμετρο, αλλά θα έχουμε όριο ανά φορτηγό, ανά τόνο δηλαδή. Πέντε, πέντε χρόνια δουλεύαμε πάνω σε μία πρόταση και τώρα ξαφνικά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Τέσσερα χρόνια παλεύεις για κάτι και τελικά έρχεται κάποιος και σου λέει ε, και τα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους και τα φορτηγά κάτω από 3,5 τόνους πρέπει να έχουν ταχογράφο. Η διαφορά ποια είναι? Καμία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι παραδείγματα τα οποία είναι τρανταχτά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε κάτι. Εγώ ήμουνα ε, στο έξι, χρόνια υπουργό στο Υπουργείο Ιστορικών, ήμουνα στην Καγκελαρία, έχω δει όλες τις μορφές της γραφειοκρατίας. Αλλά ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι αυτό που είδα στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα μάλιστα, πώς δηλαδή τόσο κουραστικά και αργά κινούνται τα γρανάζια και πόσο περιφερειακή χρειά έχουν όλα. Πραγματικά αν δεν αγαπάει κανείς τόσο πολύ την Ευρώπη μπορεί να τα παρατήσει και να φύγει. Φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε, ένα νέο, έχουμε θέσει ένα νέο στόχο πια, που νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον για σας. Ως βουλευτές, βεβαίως, εσείς ε, κατηγορείστε πολλές φορές για γραφειοκρατία και γραφειοκρατικά προβλήματα από τους ε, ε, ψηφοφόρους σας. Φρόντισα να μετρηθεί για τη Γερμανία, υποθέτω ότι μπορεί να γίνει και για τις υπόλοιπες χώρες, πόσες νομικές εντολές υπάρχουν για τον Γερμανό πολίτη τα τελευταία πέντε χρόνια. Πόσες καινούργιες νομικές διατάξεις έχουν προκύψει. Μιλούμε για έναν αριθμό 120.000 νέων νομικών διατάξεων τα τελευταία πέντε χρόνια για τους πολίτες της Γερμανίας. Το ίδιο θα ισχύει και για τους πολίτες Ιταλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, παντού. Μάλιστα εγώ εξεπλάγει για το πόσες, πόσα κίνητρα έρχονται από τις Βρυξέλλες. Πάνω από, πάνω από το 25% ε, συγγνώμη, το, πάνω από το 58% της ε, καθημερινής εργασίας έρχεται, προκύπτει από εντολές των Βρυξελών. Σαν να είναι οι Βρυξέλλες πιο σημαντικές από όσο οι χώρες. Δηλαδή παρεμβαίνουν πολύ περισσότερο οι Βρυξέλλες στις διάφορες χώρες από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Και μάλιστα πάντα έλεγα στον πρόεδρο δεν ξέρω κανένα πολιτικό επίπεδο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο αδικαιολόγητα κατηγορείται ή ε, ακούει διάφορες προσβολές για, για τόσο αυθαίρετα ζητήματα. Για, για τα πάντα φταίει η Ευρώπη έχουμε ε, ερευνήσει 77 διαφορετικές περιπτώσεις, 77 διαφορετικές οδηγίες για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες. Και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα, και μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αυτά, καταλήγουμε λοιπόν στο αποτέλεσμα ότι έπρεπε τα εθνικά κοινοβούλια να συζητήσουν μαζί σας το ότι ένα τρίτο της γραφειοκρατίας έρχεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ένα τρίτο, δηλαδή περίπου ε, περίπου 40 δις ευρώ ε, επιβάρυνση προκύπτει για την, από την μη επαρκή ή αποτελεσματική ε, εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Εγώ πήγα στην Επιτροπή Οικονομικών του, της Ανοβουλής της Γερμανίας, πήγα στη Σκανδιναβία, πήγα στην Αυστρία, γιατί πρέπει πραγματικά να συζητήσει κανείς. Γιατί χρειάζονται τόσα, ε, για τόσες διατάξεις για, ε, για, το για, για το ενοχικό δίκαιο. Γιατί χρειάζονται τόσες πολλές μέρες για να ληφθεί μια απόφαση. Η Μάλτα, ας πούμε, χρειάζεται 241 ημέρες για να εφαρμόσουν μια απόφαση. Τα έξοδα των, ε, της κυβέρνησης για τις δημόσιες προμήθειες ε, έχουν, έχουν να κάνουν με το πόσες μέρες χρειάζεται μια κυβέρνηση για να εφαρμόσει κάτι. Η Μάλτα χρειάζεται 22 μέρες, ας πούμε, και άλλες χώρε πολύ περισσότερο. Βεβαίω το θέμα αυτό έχει να κάνει και με το πόσο αργή ή γρήγορη είναι μια κυβέρνηση, αλλά από τα, από τα 27 κράτη-μέλη πάντα ε, υπάρχει κριτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν λαμβάνει κανένα υπόψη ε, το θέμα αυτό ότι κάπου αυτή η γραφειοκρατία η ευρωπαϊκή προφανώς κάπου κολλάει στο, στα εθνικά γρανάζια. Πάντα η κριτική είναι προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί και εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης και εντός του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, στην Ιστονία ένας νόμος απαγορεύει την ε, ηλεκτρονική μεταβίβαση κάποιων εκθέσεων. Στην Πορτογαλία πρέπει οι ε, διαγωνισμοί να βγαίνουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Στην ε, Πορτογαλία πάνω από 75% έχουν καλύψει την ηλεκτρονική, καλύπτεται ηλεκτρονικά η όλη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα πρέπει να υπάρχει μια βάση για να ξέρει κανείς πώς εφαρμόζει τελικά η κάθε χώρα αυτό που τη ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό, με τον Υπουργό Μεταφορών και του είπα «Πες μου, το Στουτγκάρδι 21 είναι μια, ένας σιδηρόδρομος, τον έχουμε, τον έχουμε προγραμματίσει, ε, θα γίνει από οποιουσδήποτε ε, εργαζόμενους και ο Πέτερ μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, ε, θα βάλουμε την, ε, θα συγκρίνουμε, θα πάρουμε μια ανάλυση, θα συγκρίνουμε το πώς είναι η κάθε διαδικασία σε κάθε χώρα. Τέσσερα εβδομάδες έρχεται και μου λέει άδειασα εγώ το, το σιρτάρι μου, είδα τις, τις αλλά δεν έχω αποτέλεσμα γιατί δεν μπόρεσα να συγκρίνω πώς λειτουργούν οι διάφορες διοικήσεις και αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να, να καταλήξουμε σε ένα σημείο. Πρέπει οι διάφορες διοικήσεις να ανταλλάσσουν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα όλες αυτές τις, ανα, τις αναγκαίες ε, λεπτομέρειες και τα δεδομένα που χρειάζονται. Δεν θέλω να μπω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μια τελευταία παρατήρηση θέλω να την κάνω. Πρέπει να πω, ειλικρινώς ότι έχουμε έναν Πορτογάλο ως πρόεδρο της Κομισιόν. Με την ε, σοσιαλοποίηση της ε, ε, Πορτογαλίας θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ενεργός, Παρόλο που το πρόβλημα βεβαίως στην Πορτογαλία τη γραφειοκρατία δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι όντως στην Κομισιόν τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αλλαγή νοοτροπία. Και εγώ αυτό το βλέπω και στι διάφορε διαπραγματεύσει, συζητήσει, διαβουλεύσεις που έχω με τι γενικέ διευθύνσει. Πριν από 10 χρόνια. Δεν είχε κανεί υπόψη του ότι μια ρύθμιση που είναι σημαντική ας πούμε, για το περιβάλλον ή για την προστασία του καταναλωτή ή για το εργατικό δίκαιο θα μπορούσε να έχει αρνητικέ συνέπειε για άλλου τομεί. Δηλαδή αυτό το collateral damage που λέμε σκεφτείτε τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση, όχι μόνο για τον στενό τομέα που αφορά, αλλά ποιες συνέπειες μπορεί να έχει και σε άλλους τομείς. Δηλαδή η αξιολόγηση επιπτώσεων στην Κομισιόν θα πρέπει να ληφθεί πολύ πιο σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να γίνεται πολύ πιο σοβαρά πολύ πιο σοβαρά πόσο γίνεται σε πολλές εθνικές διοικησει. Εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με, τους 27, με τις διοικήσεις των 27 κρατών μελών για την μείωση της γραφειοκρατίας. Σε κάθε χώρα προφανώς υπάρχει μια ομάδα ή ένας, ένα μεμονωμένο άτομο που προφανώς έχει διαφορετική άποψη. Αλλά χαίρομαι που ο κύριο Βίλε έχει λάβει μια δική του ε, κατεύθυνση στο θέμα αυτό για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Γιατί νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλάζουν πάρα πολλά στην ε, αντιμετώπιση της Κομισιόν. Η Κομισιόν κάνει την αξιολόγηση επιπτώσεων, αλλά το Κοινοβούλιο και κυρίω το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει αξιολόγηση επιπτώσεων. Αν τώρα το Κοινοβούλιο και με βάση την έκθεση Νίμπλερ πάει και πει ε, και ασχοληθεί με 30 ας πούμε, νέους εργαζόμενους ε, και κάνει την αξιολόγηση επιπτώσεων, θα πρέπει και ο κύριος Φαν να ασχοληθεί με το τι κάνει το δικό του ε, θεσμικό όργανο και πώς μπορεί αυτός να κάνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων. Δηλαδή κάτι κινείται αλλά πολύ αργά προς τα μπρος. Θα πρέπει να υπάρξει ε, μείωση λοιπόν της γραφειοκρατίας και από την Κομισιόν και, για το, και το Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Συνολικά όμως νομίζω ότι αν δεν έχουμε τόσο υψηλές ε, απαιτήσει, θα τα, θα, τα, θα τα καταφέρουμε νομίζω. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σκεπτικοί οι πολίτες μας σήμερα. Αν ρωτήσει κανένας κάποιον ε, στην Ευρώπη είσαι υπέρ της ε, γραφειοκρατίας ή κατά, θα σου πει κατά, προφανώς. Αλλά συγκεκριμένα ο κάθε ένας θέλει και μια ασφάλεια. Και για κάθε μέτρο, για κάθε αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε και που επιβαρύνει όμως τους πολίτες, προφανώς ξεκινάει όλη η γραφειοκρατική διαδικασία. Έχουμε και 27 κοινοβούλια Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε περιφερειακά κοινοβούλια, έχουμε 27 κυβερνήσει. και προφανώ όλοι αυτοί σκέφτονται για το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών. Και βεβαίω όλοι αυτό προσπαθούν να το κάνουν με νέε νομοθετικέ ρυθμίσει. Δεν έχω δει κανέναν μέχρι στιγμή να λέει να κάνουμε λιγότερε νομοθετικέ ρυθμίσει για να εξασφαλίσουμε του πολίτε. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει απαιτεί πολλή γραφειοκρατία επιβάλλοντα και άλλη γραφειοκρατία. Γιατί μετά κατηγορούνται οι πολιτικοί ότι προσπαθούν να καταλύσουν την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτε. Αυτά από μένα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, προσπάθησα και εγώ να σας δώσω έτσι ε, λίγη τροφή για σκέψη. Ε, παρακαλώ όμως να κρατήσετε τα, στο, στο νου σας το θέμα αυτό και να το προωθήσετε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Δόκτωρ Στόιμπερ για την παρουσίασή σας στην σημερινή μα συνεδρίαση βρήκα και εγώ ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να μειώσει τα έξοδα. Μπορεί κανείς να βρει πολλά παραδείγματα για πολλά για πολλά άσκοπα έξοδα, αλλά κανένα δεν είναι τόσο παράλογο όσο το που πρέπει να βρίσκεται ο τείχος ενός νεκροταφείου. Να δώσουμε τώρα λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους για την παρουσίαση αυτή. Παρακαλώ, 1,5 ε, λεπτό ο καθένα, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε και την, ε, και την ε, ψηφοφορία. Η κυρία Γκρέσλε πρώτα και μετά η κυρία Γιάλα Σέντερ. Να πω εγώ από το ΕΛΚ ότι πώς μπορώ, αυτή η έκθεση είναι νομίζω η καλύτερη που έχουμε διαβάσει για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την Ευρώπη. Κυρίω γιατί πραγματικά μιλά για ένα πρόβλημα το οποίο το θεωρούν όλοι πρόβλημα. Πώς δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε και την ε, ε, εφαρμογή των νόμων αλλά και χωρίς να επιβαρύνουμε ε, τους πολίτες. Είναι δύο κόσμοι που πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδυαστούν. Γιατί προφανώ υπάρχουν πολλέ παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θέλω να. Προφανώ και εμεί θέλουμε να συνεχίσετε την δουλειά σα. Θέλουμε περισσότερε ευκαιρίε για να συζητούμε τα θέματα αυτά το, αυτό που λείπει πάντα είναι κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες ιδέες. Έχει γραφτεί πάρα πολύ ωραία αυτή η, ε, αυτή έκθεση, δεν έχει αυτό το, τη γλώσσα την ευρωπαϊκή. ασχολείται ακριβώς με την ουσία των πραγμάτων. Είναι λοιπόν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Είπατε ότι 85% ε, επιστρέφει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλω να μας δώσετε κάποια στατιστικά από αυτά που είπατε. Και εγώ κάνω κάποιες μετρήσεις για την ομάδα των χριστιανοδημοκρατών και νομίζω ότι περίπου το 1 τρίτο της, ε, των δαπανών ε, εκτελούνται. Οπότε θα ήταν καλό να λάβουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και ίσως από την Κομισιόν θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε καλύτερα την κατάσταση. πολλά κράτη-μέλη ουσιαστικά προσπαθούν να μπουν μείωση της, ε, ε, της ε, γραφειοκρατίας, αλλά απ' την άλλη δεν θέλουν να αναλάβουν και την ευθύνη. Δεν θέλουν να υπάρχει λογοδοσία. Δεν θέλουν να του ρωτάει κανείς πού τα δώσετε τα λεφτά αυτά. Ναι, είναι καλό να πουλάμε την μείωση τη γραφειοκρατίας, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερη λογοδοσία. Βεβαίω καλύτερη λογοδοσία από ό,τι είχαμε μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να συλλέξουμε λίγο τι ε, παρεμβάσει. Η κυρία Γιάλα Σέντερ και μετά η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στόιμπερ για την παρουσίασή του και για την προσήλωση που δείχνει σε αυτή τη δουλειά. Να σχολιάσω το εξή μόνον με επηρεάζει άμεσα το θέμα του ψηφιακού ταχογράφου. Ε, δεν λάβατε υπόψη, ενδεχομένω κύριε Στόιμπερ, τις οργανώσεις ε, των θυμάτων ε, ε, στους αυτοκινητόδρομους αυτοκινητικών δυστυχημάτων, διότι σίγουρα αυτοί έχουν πληγεί περισσότερο ε, τα μικρά φορτηγά να διανύουν 150 χιλιόμετρα χωρίς ταχογράφο, οκ, okay, αλλά ε, μπορώ να σας πω ότι ανάμεσα στο, στην Αλκαλά Δενάρης και στη Μαδρίτη που είναι μια απόσταση 50 χιλιόμετρων θα συμβούν πάρα πολλά ατυχήματα ε, εξαιτίας τέτοιων φορτηγών και τέτοιων οδηγών που δεν ξεκουράζονται όπως πρέπει και όταν πρέπει. Να σας ε, ρωτήσω το εξής για τα συμπεράσματά σας. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα. Ε, πολύ δε περισσότερο εξαιτία του ότι εγώ έχω και συγκεκριμένες ευθύνες ε, στην Ισπανία σε τοπικό επίπεδο. Ε, τα αποκεντρωμένα κράτη, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, ε, έχουν τρία επίπεδα ε, νομοθετικής εξουσίας. Πολύ συχνά σε αυτή την κλίμακα ε, εφαρμογής σε τρία διαφορετικά επίπεδα ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα. Ε, πώς, ποιες ήταν οι καλύτερες πρακτικές να το βελτιώσουμε αυτό. Δεύτερον, η ενημέρωση του κοινού, η επικοινωνία. Πώς είναι δυνατόν να δείξουμε στο κοινό ότι οι Βρυξέλλες είναι σημαντικές και ότι δεν είμαστε τόσο κακοί πάντοτε ή τόσο ανίκανοι διοικητικά. Η ομάδα υψηλού επίπεδου πώς πιστεύει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας στρατηγική. Τρίτον, ε, μία πτυχή είναι η μείωση των, της νομοθεσίας, αλλά όχι βέβαια να καταργήσουμε και τους σημαντικούς. Γιατί είδαμε τώρα στην κρίση που, ότι υπήρχαν κάποιοι κανόνες που δεν εφαρμοζόντουσαν και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε κρίση. Θα πρέπει να ισορροπήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Στόιμπερ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μια παρατήρηση ο πρώην Πρωθυπουργό ε, της ε, Βαβαρίας ε, είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών στο Συμβούλιο και αυτό είναι ένας λόγος γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά γιατί εγώ είμαι εδώ στο, σε αυτή την ομάδα, την Επιτροπή του Κοινοβουλίου ένα μήνα και βλέπω τα, τα πράγματα έτσι ίσως λίγο διαφορετικά για το τι είναι τελικά σωστό. Ε, πιο αξιόπιστο ε, ομόλογο από εσά, συνομιλητή από εσά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Πρέπει να δούμε αυτά τα λάθη της εφαρμογής ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Πρέπει να έχουμε και τη βοήθεια βέβαια του ελεγκτικού συνεδρίου. Είπατε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκοι οι ε, κανόνες που διέπουν τις δημόσιες προμήθειες. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να υποστούν μια μεταρρύθμιση. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε μια μοναδική ευκαιρία για, με την συνεργασία και την, ε, με τη δική σας την ομάδα υψηλού επίπεδου. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή ε, ευκαιρία να κάνουμε όλοι ό,τι, πρέπει για, τις, για τους ε, κανόνε για τι δημόσιες προμήθειε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή όσων θέλουν να ε, βγάλουν και κάποια χρήματα από τις δημόσιες προμήθειε. Και επίση μπορούμε να βοηθήσουμε και την Ευρώπη γιατί όταν θα κάνουμε του κανόνε πιο απλούς προφανώ θα γίνουν και τα λάθη πιο μικρά και πιο λίγα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία συνεργασία και θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να κάνουμε πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η επόμενη κυρία Χολμάιερ. Ήθελα να πω στην αρχή, κύριε Πρόεδρε της ομάδας υψηλού επίπεδου, κύριε Στόιμπερ, αυτό το θέμα με τους ταχογράφους Νομίζω έχει, έχουν υπάρξει πάρα πολλέ ε, παρεξηγήσει ε, γύρω από αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ τη ε, αλλαγή των κανόνων οι ε, εργάτες ή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που ε, παλεύουν απέναντι στην κρίση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορούν να δώσουν ένα, ένα μήνυμα, να δώσουν το πράσινο φως για την μείωση αυτής της γραφειοκρατίας. Το ερώτημά μου προς την δική σας ομάδα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί η ομάδα σας να δώσει κάτι πιο δεσμευτικό από τις απλές ε, προτάσεις ή συστάσεις έτσι ώστε να προσπαθήσει κανείς να βελτιώσει τα πράγματα και να ρυθμίσει καλύτερα και πιο ενιαία όλους αυτούς τους κανόνες αντί να πρέπει να έρθει σε επαφή με 25 διαφορετικές υπηρεσίες που μπορεί να έχουν ε, τελείως διαφορετικές απόψεις, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει και τους ελέγχους. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον, να, να ζητήσω μάλλον από, τους, ε, από τον κύριο Σίμψον και την Επιτροπή του να μιλήσει ίσως γιατί ο κύριο Στόιμπερ είναι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από του δύο επόμενου ομιλητέ να μην πάρουν το λόγο και να αφήσουμε τον κύριο Στόιμπερ να μα απαντήσει. Μήπω μπορείτε κύριε Στόιμπερ να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας τέθηκαν. Ξεκινώντας από το τέλος, την κυρία Χολμάιερ. Να πω το εξή. Να ξεκαθαρίσω λίγο τι έχουμε κάνει, έτσι ώστε να καταλάβετε κι εσείς τι γίνεται. Εγώ έχω γράψει επιστολές σε όλους τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, σε 27 δηλαδή. Και ε, αυτό είναι και το ερώτημα του κύριου Γκάιερ. Του ζήτησα Δώστε μου ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Κάτι που έχετε εφαρμόσει πάρα πολύ καλά. Δεν του ζήτησα αρνητικά παραδείγματα γιατί δεν θα είχα τίποτα. Και 27 λοιπόν αρχηγοί μου ζήτησαν, μου έστειλαν παραδείγματα για το πόσο ωραία έχουν εφαρμόσει το ένα και το άλλο. Κύριε Γκάιερ λοιπόν, όταν κάποιο είναι ο καλύτερο, υπάρχουν και ε, προφανώ κάποιε χώρε που δεν είναι από του πρώτου, είναι τελευταίε. Οπότε στα εθνικά τους κοινοβούλια, στα εθνικά, στα εθνικά κοινοβούλια, πρέπει να τεθεί, να το ερώτημα, εσείς οι Γάλλοι ας πούμε, γιατί δεν είσαστε καλύτεροι σε αυτό. Η κυβέρνηση τι κάνει. Ελπίζω να μπορέσουμε λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά Νομίζω ότι στην Αγγλία κάτι τέτοιο γίνεται και στις σκανδιναβικέ χώρες επίσης κάτι παρόμοιο γίνεται, στη Γερμανία γίνεται και στις χώρες Μπενελούξ επίσης. Αλλά υπάρχει, έχει γίνει έτσι ένα μικρό βήμα, δημιουργείται μια νέα κουλτούρα. Και αγαπητή Μόνικα, έχουμε καταλόγους για την εφαρμογή. Βλέπει εδώ, του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έχουμε δέκα περιπτώσεις, δεν θέλω να σας τις ε, διαβάσω, αλλά, ε, δείτε κυρίες ε, και κύριοι της κυβέρνησης στην Ρώμη πώς μπορείτε σε αυτό τον τομέα να βρείτε μια βέλτιστη πρακτική. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα, τα στοιχεία. Ελπίζω να, να ξεκαθαρίζονται έτσι λιγάκι τα πράγματα, γιατί το θέμα του δικαίου, των ηχικού, δεν το κατακρίνω, αλλά Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς το ένα συγκρούεται με το άλλο τελικά, λόγω ακριβώς της γραφειοκρατίας. Στη μία χώρα, ας πούμε, εφαρμόζεται έτσι το, το, το δίκαιο, στην άλλη χώρα εφαρμόζεται αλλιώς. Προφανώς αυτό έχει επιπτώσεις και στην εσωτερική αγορά. Κυρία Γκάιερ, να πω ότι υπάρχουν και περιφερειακά συμφέροντα. Ε, Βέβαια πάντα το θέμα είναι οπτικής γωνίας. Ε, προφανώς ξέρω ποια είναι τα ε, περιφερειακά ε, συμφέροντα. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της επικουρικότητας. Και σας λέω σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το εμπορικό της ισοζύγιο και οι αλλαγές και ας πούμε η υποχρέωση δημοσίευσης για μικρές επιχειρήσεις είναι πραγματικά λυπηρό και, στην, ε, και στο ε, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ήμουν εκεί, ήμουν παρόν και ξαφνικά ένα Πορτογάλος ε, έρχεται με το πρόβλημα τη πορτογαλία, μετά η Αυστραλία λέει όχι εμεί δεν έχουμε πρόβλημα, η Πολωνία λέει ναι και εμεί έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Γίνεται ένα χάο. Και κατά τη δική μου άποψη, σε τέτοια πράγματα η Κομισιόν πρέπει να παρεμβαίνει πολύ πιο δυναμικά και να λέει ναι, ωραία, υπάρχει ένα περιφερειακό συμφέρον εδώ, αλλά υπάρχει και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και αυτό θα πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Νομίζω ότι ε, εμείς ε, οι δύο συμφωνούμε σε αυτό. Το θέμα των ε, δημοσίων προμηθειών και ο τρόπος με τις, ε, που θα εφαρμοστεί η σχετική οδηγία θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει κάποιο στη Μάλτα να, ε, να, να, να, σκεφτεί λίγο γιατί ας πούμε στην, ε, στο αντίστοιχο τομέα στην Λιθουανία χρειάζονται τόσο λίγα χρήματα. Θα είναι λοιπόν αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Τώρα για την κυρία Γιάλα Σέντερ. Πάλι φτάνουμε στο ερώτημα ελευθερία ή ασφάλεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προσπερνάμε αρκετά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να, α, να δέσουμε ένα παντελόνι με μία ζώνη. Όταν ξέρετε ότι ίσως ε, ο τρόπος με τον οποίο δένετε τη ζώνη να καταστρέψει τη ζώνη, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Για να μπορέσετε δηλαδή να φορέσετε και το παντελόνι σα, για να μην σα πέσει, να δέσετε σωστά τη ζώνη, να φορέσετε και το πουκαμισό σα. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν. Κάτι παρόμοιο κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι, εντάξει, στη Μαδρίτη ή οπουδήποτε αλλού ε, μπορεί να υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, κατευθυντήριες γραμμές, πάρα, πολλά, πάρα πολλοί μεταφορείς, πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Αλλά αυτοί οι ταχογράφοι αφορούν τους επαγγελματίες οδηγούς. Αυτούς δηλαδή που όντως ταξιδεύουν 50 ώρες τη βδομάδα. Αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε, να μην οδηγούν πάνω από τις ώρες αυτές, να έχουν ώρα ξεκούρασης. Αλλά πρέπει να πω πρέπει να το δούμε ακριβώς, πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό. Το πουκάμισο, το παντελόνι και τη ζώνη, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα τρία από κοινού για να συνδυάσουμε όλα αυτά. Δεν μιλάμε για ανθρώπου που οδηγούν πάρα πολύ λίγε ώρε. Δεν, δεν χρειάζονται όλοι ταχογράφο. Αυτό είναι υπερβολική απέτηση. Θα μπορούσα ώρε να σα μιλάω για αυτά. Αλλά για τα παιδικά παιχνίδια, α πούμε, και τη σχετική οδηγία. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που έχει γίνει. Αν θέλετε να θέσετε σε εμπορία ένα παιχνίδι σήμερα, πρέπει είτε να πάτε στο Λονδίνο ή πρέπει να, φέρ, βρείτε 100 παιδιά για κάποιους μήνες, τα οποία παιδιά πρέπει να πάρουν ας αυτό το παιχνίδι και να παίξουν το, ε, ή το, ε, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλετε να θέσετε σε εμπορία. Και αν ε, δεν το χρησιμοποιήσουν σωστά, τότε έχει αποτύχει το, το προϊόν σας. Ναι, ωραία, μπορεί η, ε, η γραφειοκρατία, ας πούμε, για τα ε, για τα βεγγαλικά να είναι ε, υπερβολική, αλλά αν μπορέσουμε να ε, σώσουμε και από τα, ένα, έστω και ένα παιδί από αυτά, λόγω ακριβώ γραφειοκρατία, αυτό είναι καλό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μεν κάποιε ασφαλιστικέ εκλίδε, αλλά να έχουμε και ε, μια αλφα ευελιξία. Εγώ απλώ θέλω να σα πω ότι πρέπει να έχουμε έτσι ένα περιθώριο και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη ο καθένας προσωπικά ανάμεσα σε αυτή την ε, ασφάλεια που θέλουμε να εξασφαλίσουμε αλλά και την ελευθερία που θέλουμε να έχουμε. Και ναι, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή είναι σωστό κυρία Γκρέσλε αυτό που λέτε αλλά νομίζω ότι εδώ στο Συμβούλιο ε, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Γιατί αυτοί ακριβώ έχουν πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με το πώ εφαρμόζεται η νομοθεσία σε σχέση με την Κομισιόν και, την, και το Κοινοβούλιο. Ε, ξέρω ότι τα είπα λίγο γρήγορα, αλλά ήταν λίγο και ο χρόνο. Κάποιοι Γάλλοι συνάδελφοι μου είπαν ότι κάνω και κάτι καλό. Δεν το έχω φανταστεί, δεν το περίμενα. Ελπίζω όμω να μπορέσουμε όλοι από κοινού να προωθήσουμε το στόχο αυτό για την λιγότερη γραφειοκρατία. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που με καλέσατε. σα ευχαριστώ όλου και ό,τι καλύτερο σα εύχομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Στόιμπερ. Χαίρομαι που δεν μιλήσατε για του φιλελεύθερου. Ίσως να μην αξίζουν τον έπαινό σας να πω, δεν ξέρω πώς να το εκλάβω αλλά και εγώ ως ε, φιλελεύθερος πρέπει να πω ότι οι ιδέες αυτές ε, ότι πρέπει δηλαδή να προσανατολιστούμε προ προς, τους, ε, προς καλύτερες πρακτικές για το μέλλον θα μπορούσε όντω να αποτελέσει μια νέα προσέγγιση για, τους, για την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμού. Να μην δούμε δηλαδή μόνο ποιο κάνει τα περισσότερα λάθη αλλά, λάθη, αλλά να δούμε και τι λειτουργεί καλύτερα. Να προσανατολιστούμε λοιπόν προς τους καλύτερους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ανήκετε όντω στου καλύτερους που έχουμε καλέσει στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ ζωντανή συζήτηση που κάναμε σήμερα. Ε, και ήμουν και εγώ και, στην, ε, και στους φιλελεύθερους αρκετά. Μάλιστα ήταν οι πιο εντατικές και οι πιο ζωντανές συζητήσεις που έκανα ήταν μαζί με φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Äh, λοιπόν, αποχαιρετούμε τον κύριο Στόιμπερ. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη στην εφαρμογή των προτάσεών του για την μείωση της γραφειοκρατίας. Όσοι είναι υπεύθυνοι από την ΙΜΚΟ για τα παιδικά παιχνίδια, τους ευχηστώ την προσοχή. Äh, λοιπόν, πάμε. Να πω μάλλον ότι θα επανέλθουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης μετά από αυτή την αλλαγή ε, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ε, ειδική έκθεση νούμερο 12 Εισηγείται η κυρία Αντρέασεν. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Yeah. Okay. Ähm, ähm, wir kommen äh, zur Abstimmung. Ψηφίζουμε λοιπόν. Σημείο 4. Ε, για την ε, ειδική έκθεση 2000, υπαριθμών 12, 2011. Λοιπόν, παράγραφος 3. Τροπολογία 2. Είναι σε γέλα σέντερ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι, δεν έχετε ψηφίσει όλοι. Α, δεν έχει κλείσει ακόμα η ψηφοφορία. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι σωστό. Απορρίπτεται. Μάλλον δεν έχουν ψηφίσει όλοι όμως παρόλα αυτά. Έχουν, έχετε βάλει όλοι τις κάρτες σας, έχετε... Έχει κανείς αντίρρηση με το αποτέλεσμα, όχι. Γιένς Γκάιερ, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεν ήταν σαφέ. Υπέρ παρακαλώ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, γκρίνεται. Τροπολογία 5 καταπίπτει. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Α, η 6, συγγνώμη, η 6 καταπίπτει. Η 8... Ε, α, συγγνώμη, ναι, η 6 υπάρχει υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ, 9, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 καταπίπτει. Τροπολογία 10. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Για τη 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη συμβαστική 1 συμβαστική 1 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Amendment number 1. Hat jeder abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Κάποιο έχει ξεχάσει την κάρτα του. Α, κάποιο άφησε την κάρτα του στο μηχανηματάκι. Εντάξει, κλείνουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Εγκρίνεται. Η 15 καταπίπτει, η 16 καταπίπτει, η 17. Ψηφίζουμε τη 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τροπολογία 18. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Moment. Ja, es nur 17 sind anwesend. Okay, dann. Äh... Κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 αποσύρεται. 25 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 ε, κατά αν υιοθετηθεί 23, αλλά 23 αποσύρθηκε. Η 25... Λοιπόν, άρα αυτές καταπίπτουν. Πάμε στην ΠΕΣ 1. 1. Η επόμενη που θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ΠΕΣ 1. Hat jeder abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πεσ 2. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πεσ 3. Υπέρ. Κακά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πεσ 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέντε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες έξι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πες έξι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε την ΠΕΣ 7. Hat jeder abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ισοπαλία στις ψήφους. ΠΕΣ 8. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πες 9. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάλι ισοπαλία. Πες 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα. Την ΠΕΣ 10. Δεν είναι απόλυτα σαφέ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ΠΕΣ 10. Πέρας ψηφοφορια εγκρίνεται. ΠΕΣ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. ΠΕΣ 12. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έκθεση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας φορείας. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στην κυρία Αντρέασεν. Πάμε στην επόμενη έκθεση. Τάμας Deutsch. Έκθεση Τάμας Deutsch. Ψηφοφορία για την ε, τροπολογία στην παράγραφο 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ να το δούμε. Ψηφίζουμε τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άφετ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα unblock. 2 με 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης του Τάμας Deutsch. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο των ψηφοφοριών. Πολύ ωραία. Um, colleagues, dear colleagues, uh, please um, Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της μερίσιας διάταξης και να δούμε από εκεί και πέρα την απολογή του Συμβουλίου, διότι είναι εδώ τα μέλη του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να φύγετε. Are you there tomorrow? Are you here tomorrow? Θα είστε εδώ αύριο. Ωραία. Λοιπόν, αναβάλλεται η απαλλαγή του Συμβουλίου για αύριο. Αύριο το πρωί θα γίνει το σημείο 6. Το 7. Μήπω θα μπορούσε να είναι το πρώτο σημείο, διότι έχω κάνει και εγώ το πρόγραμμά μου και δεν θα μπορώ να είμαι εδώ αργότερα. First point tomorrow. Ωραία, πρώτο πρώτο σημείο αύριο το πρωί. Πάμε στο σημείο 8. Σημείο 8. Ειδική Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία. Πέτυχε η Κομισιόν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Ο συνάδελφος Γκάιαρ είναι ο εισηγητής. Δεν ξέρω αν ο εισηγητή θέλει πρώτα το λόγο ή να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον ελεκτικό συνέδριο. Πρώτο εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Λαζάρου και όλους τους συνεργάτες. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η να δωσουμε κατευθειαν το λογο στο ελεκτικο συνεδριο πρωτο εισηγητη ευχαριστω προεδρε Καταρχά να ευχαριστησω τον κυριο λαζαρου και ολους τους συνεργατες πραγματικα ηταν πολυ ενδιαφερουσα η εργασια που έγινε. Και θα ήθελα πραγματικά να επενέσω όλους τους συναδέλφους. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι τα λάθη που γίνονται στην περιφερειακή πολιτική είναι το σημείο που πάντα ανακύπτει και μας δημιουργεί προβλήματα στις αιτήσεις διαδικασίες απαλλαγής. Και το θέμα είναι αν ε, τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση λειτουργούν σωστά και πώς ε, αντιδράει η Κομισιόν αν ε, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό σημείο για να δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα λάθη που γίνονται στην περιφερειακή πολιτική. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει 40 περιφερειακά προγράμματα στα, τα οποία έχει ερευνήσει. Έχει θέσει τρία ερωτήματα. Αν έχει δηλαδή κάνει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα η Κομισιόν, αν έχει ε, ε, φροντίσει να γίνει άμεσα αυτή η διόρθωση και αν έχει ε, εξασφαλίσει την, σωστή ασφα... την επαρκή ασφάλεια για, το... για την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αληφθεί. Το αποτελέσματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι η, η διάρκεια α, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή το πόσο κρατάει, πόσο παίρνει η, όλη η διαδικασία αυτής διόρθωσης των ε, λαθών στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, ερευνήθηκαν προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου ε, για 27 μήνες. Ε, για την ε, Γενική Διεύθυνση ε, Ρέγγιο 32 μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μου ζητήθηκε να μιλήσω για την ευθύνη των κρατών μελών και να την τονίσω. Γιατί ούτως ή άλλως τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να λάβουν τα διορθωτικά μέτρα που επιβάλλει η αλλως τα κρατημέλη ειναι αυτα που πρεπει να λαβουν τα διορθωτικα μετρα που επιβαλλει η κομισιον και προφανώς έχουν και αυτά συνευθύνη. Οπότε πρέπει λοιπόν να δούμε γενικώ τι γίνεται και ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε στο μέλλον για να μειώσουμε την διάρκεια αυτή τη περίοδου που, παίρνει, που διαρκεί αυτή η διόρθωση των μέτρων. Επίσης σημαντικό είναι το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η έκθεση πριν το πρόγραμμα δράσης της ε, Κομισιόν και της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Πολιτικής, πριν το 2008 δηλαδή, πριν το σχέδιο δράσης αυτό, πολλά από τα λάθη και τις ελλείψεις που παρατήρησε το ελεκτικό συνέδριο τα διαχειρίστηκε η Κομισιόν. Οπότε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου Ε, δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα αυτά, τα λάθη αυτά. Περιλαμβάνονται μόνο τα λάθη τα οποία δεν έχουν διορθωθεί και τα οποία έχουν, ε, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό θα πρέπει ε, στη διαδικασία απαλλαγή να δούμε όντω αν αυτό που λέει η Κομισιόν ότι έχει κάνει για να καλύψει τι λήψει και τα λάθη, να όντω έχει εφαρμοστεί σε ένα βαθμό που να μπορούμε να πούμε ότι μα ικανοποιεί. Δεύτερο σημείο. Δεύτερο ερώτημα που έθεσε το ελεκτικό συνέδριο. Η Κομισιόν έχει δημιουργήσει την απαραίτητη ασφάλεια ώστε αυτά τα μέτρα που ζητούνται να ληφθούν έχουν ε, ληφθεί επαρκώς ε, για την, ε, ώστε να μπορούν τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της Κομισιόν να λειτουργούν σωστά. Άρα το έλεγχος που έκανε η Κομισιόν ήταν επαρκής αν έγινε αξιολόγηση επίσης της, από την Κομισιόν των διαφόρων μέτρων που έλαβαν οι διάφορες εθνικές αρχές. Και, αυτό, και εδώ πάλι η έρευνα έγινε πριν το πρόγραμμα δράσης. Ε, το ηλεκτρικό συνέδριο δεν είναι ικανοποιημένο ή τέλο πάντων δεν ήταν ικανοποιημένο τότε. Σε 78% των περιπτώσεων η Κομισιόν ε, μετά την πρώτη αξιολόγηση ε, συνεπειών μπορούσε να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα και αυτό δεν ήταν θετικό. Και αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ ανησυχητικό γιατί αν δούμε τι σημαίνει αυτό σε πολιτικού όρου, σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν, κράτη, έχουν συστήματα διαχείριση και ελέγχων που δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα κράτη-μέλη διαπιστώνουν ότι δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, χρειάζονται βοήθεια, αλλά στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η Κομισιόν έρχεται μετά την αξιολόγηση των συνεπειών να πει ότι δεν ήταν επαρκής η, ε, η λειτουργία των συστημάτων. Οπότε πρέπει να δει και η Κομισιόν την ευθύνη που έχει για το πώ βελτιώνονται τα συστήματα διαχείριση και έλεγχου. Οπότε δεν είναι αξιοπεριεργό που τα λάθη δεν μειώνονται. Επίση, τα κράτη-μέλη δίνουν πολύ λίγα δεδομένα, πολύ λίγε πληροφορίε στην Κομισιόν και η Κομισιόν ε, επαφίεται σε πληροφορίε των κρατών μελών, χωρί όμω να, να ε, εξετάζει την αξιοπιστία αυτών των ε, πληροφοριών. Και πρέπει επίση να πω αν το πρόγραμμα δράσης από το 2008 και μετά οδήγησε στο ότι αυτή η αξιοπιστία της Κομισιόν να είναι μεγαλύτερη πια. Να μπορεί δηλαδή η Κομισιόν να βασίζεται στα δεδομένα που ε, λαμβάνει από τα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, ε, θέλει να μειώσει τον αριθμό λαθών μετά από δύο χρόνια ο, μειώθηκε ο αριθμός των λαθών. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τα ιδιορθωτικά ταμεία. Το την τελευταία φορά που το, που, είδαμε, που το είδαμε είχαν αυξηθεί και πάλι τα λάθη. Εξεκολουθούν να είναι αρκετά, υψηλά, αρκετά υψηλός ο αριθμός και η τάση είναι να παραμείνει υψηλός. Και αυτό μάλιστα μένα με ανησυχεί. Αλλά πρέπει να πω πάλι, για να είμαστε δίκαιοι, ότι το επίπεδο των λαθών που καταγράφονται έγινε πάλι πριν το 2008. Ελπίζουμε ότι τα λάθη αυτά ε, που είχαμε τότε δεν θα ξαναγίνουν. Δεν θα είναι δηλαδή ο αριθμός τόσο υψηλός. από το 2008 ε, θα έπρεπε να φαίνεται ένα σημαντικός, μια, σημαντική μείωση των ε, λαθών και καλό θα ήταν να μάθουμε από την Κομισιόν πόσο σημαντικός τελικά ήταν ο αντίκτυπος των ε, διορθωτικών μέτρων για το σύνολο των λαθών. Είχαμε δύο ευκαιρίες να μειώσουμε τα λάθη. Ο ένας είναι μέσω καλύτερων ελέγχων. Κάναμε και τη συζήτηση με, με τον Στόιμπερ για το τι γίνεται με τα λάθη. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κάποια λάθη μέσω οικονομικών διορθώσεων να, να ε, διορθωθούν συνολικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το σχολιάσει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά για τον Ευρωπαίο φορολογουμένο είναι σημαντικό. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και αν έγιναν τα λάθη αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους, με, τις μεθόδους μέσω οικονομικών διορθώσεων να διορθώσει αυτά τα, τα λάθη. Το ερώτημα τώρα είναι... αν μπορούμε να μπούμε σε μια ουσιώδη συζήτηση με την Κομισιόν ως προς αυτό. Συμπέρασμα λοιπόν από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι θα πρέπει άμεσα για την περίοδο 2007-2013 να εφαρμοστούν τα διάφορα μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά την διάρκεια και την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σου σχόλια. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Λαζάρου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση υπαριθμών 3 του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 μια αξιολόγηση για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε επαρκώς τι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τα διαρθρωτικά ταμεία δράτω με τις ευκαιρίες εξ ονόματός μου και της ομάδας μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Γκάγερ και την ομάδα του για την αγαστή συνεργασία που είχαμε για την εκπόνηση της έκθεσης. Το σχέδιο έκθεσης που ετοίμασε ο εισηγητής, ο κύριος Γκάγερ, παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα της ειδική έκπαιδευσης του ελεκτικού συνεδρίου, γεγονός που μου επιτρέπει να είμαι λακωνικό στην παρουσίασή μου. Ο έλεγχο έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι ελλείψη στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 έγινε καταλήλω. Έγιναν πολλές διορθώσεις για να ε, προασπίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και σε πολλέ περιπτώσει, τα κράτη-μέλη κατάφεραν να ε, αντικαταστήσουν ε, τι παράτυπες δαπάνε ή να τι αποσύρουν. Ε, δεν είχαμε βέβαια πλήρη αποτελέσματα, διότι έπρεπε να γίνουν και κάποιες επιπλέον διαδικασίες και επιπλέον δημοσιονομικές διορθώσεις θα απαιτηθούν στο μέλλον. Χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να έχουν καλύτερα ποιοτικά συστήματα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο έλεγχος δεν ε, κάλυψε και τη διαδικασία καθάρισης, διότι είναι ακόμα εν εξελίξη μετά από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι οποίες δεν ήταν επαρκή σε όλες τις περιπτώσεις οποίες ε, διαπιστώθηκαν προβλήματα, ε, η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως δίκτυ ασφαλείας. έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι εκαθάρισης για περιορισμένο αριθμό ε, περιπτώσεων και θα πρέπει από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί στις ε, ε πληροφορίες που της δίνονται για τις εκαθαρίσεις και αυτό εκπείρας ε, δείχνει ότι οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι αρχές των κρατών μελών δεν είναι πάντα οι απόλυτα ορθές δηλώσεις ε, και αλλαγές. Θα πρέπει επίσης να γίνει σωστή αξιολόγηση του ποσοστού σφάλματος του προγράμματος όπως παρουσιάστηκε από την αρχή εκαθάρισης. Αν ε, υπερβαίνει το κατόφλι του 2% τότε θα πρέπει να γίνουν δημοσιονομικές διορθώσεις βάσει των προβολών του ποσοστού σφάλματος. Από εκεί και πέρα θα γίνουν διορθώσεις για κάποια προγράμματα κατά την εκαθάριση και τα κράτη-μέλη, όπως σας είπα προηγουμένως, μπορούν να, να αντικαταστήσουν τη δαπάνη που έχει ε, διαπιστωθεί ως μια επιλέξιμη στο παρελθόν. Αυτό γίνεται διότι τα κράτη-μέλη μπορούν να δηλώσουν δαπάνες άνω του προπολογισμού που έχει δοθεί και έτσι έχουν μια δικλίδα ασφαλείας για να διορθώσουν και να κάνουν τις απαραίτητες δημοσιονομικές διορθώσεις. Οι αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν αλλαγές ε, για τη δυνατότητα αντικατάστασης δαπανών που ε, θεωρούνται μη επιλέξιμες στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Δεδομένου ότι κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται σε ε, δινή οικονομική θέση και έχουν λάβει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα, θα πρέπει ε, να βρεθεί διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανασταλτικών μέτρων και μέτρων τα οποία γίνονται για διορθώσεις. Όπως είπε και ο κύριος Γκάγερ στο σημείο 12 του σχεδίου έκθεσης, αυτό γίνεται προ όφελο των κρατών μελών. Θα πρέπει να έχουν συστήματα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι είναι ε, οι συναλλαγέ και φυσικά ε, έχουμε και την κατάλληλη αξία για τα όσα πληρώνουμε. Και φυσικά ε, δεν θα πρέπει να κατασπατελούνται δημόσιοι ιδιωτικοί πόροι. Επομένως, διακυβεύονται και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Δεύτερον, στην περίπτωση που κάποιε δαπάνε δεν θεωρούνται επιλέξιμες από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπές και επομένω δεν επιτρέπονται, ε, θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικά ή περιφερειακά κονδύλια. Ο φορολογούμενος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ε, πλήτεται σε αυτή την περίπτωση και θα πρέπει να φροντίζουμε να είναι σωστοί οι λογαριασμοί μας. Οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ε, ε, ταμείων προβλέπουν διάφορα επίπεδα ελέγχων. Ε, καταρχάς γίνονται έλεγχοι σε πρώτο επίπεδο από τις αρχές πληρωμές ή βάση δικη τους εξουσιοδότησης και από εκεί και πέρα οι έλεγχοι σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να γίνονται από τις ελεγκτικές αρχές. Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχουμε μια βελτίωση. Οι αρχές ε, ελέγχου θα πρέπει να δίνουν αιτήσια ποσοστά σφάλματος βάσει ε, αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από στατιστική σκοπιά. Ε, αντιπροσωπευτικά δείγματα από στατιστική σκοπιά σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε προβολή των αποτελεσμάτων. Επομένω, αυτή η έλεγχο σε δεύτερο επίπεδο είναι ο τρόπο διασφάλιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω λέει και ο ίδιο ο εισηγητή, εάν και μόνο εάν αυτοί οι έλεγχοι μας δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα, από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να διασφαλίσει νομιμότητα και σωστούς λογαριασμούς και θα γίνονται δημοσιονομικές διορθώσεις βάσει του σωστού ποσοστού σφάλματος. Και τέλος, επειδή ενισχύονται σε σημαντικό βαθμό οι έλεγχοι σε δεύτερο επίπεδο, τα διάφορα επίπεδα διαστρωμάτωσης ε, ε, των ελέγχων μπορεί να επανεξεταστούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, Σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά βεβαίως υπάρχει και η έκθεση της Κομισιόν. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ντεφά 80% ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει να κάνει με τις ε, κοινέ αρμοδιότητες και βεβαίως τα διαρθρωτικά ταμεία είναι σημαντικά ως προς αυτό. Ο κύριος Ντεφά θέλει να απαντήσει σε ερωτήματα, αλλιώ να δώσουμε και τον λόγο στους συναδέλφους για να θέσουν τα ερωτήματά τους, οπότε δεν ξέρω, θέλετε κατευθείαν το λόγο, θέλετε να δώσουμε ο κύριος Ντεφά πρώτα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, πολύ σύντομα. Ε, γιατί επειδή ακριβώς συζητούμε το θέμα αυτό για το πώς βλέπουμε εμείς την έκθεση και, ένα, και θα ήθελα να θίξω και δύο σημεία που είπε ο κύριος Λαζάρου αλλά παρακαλώ να, να το κάνετε σύντομα ώστε να μπορούν να παρέμβουν και τα μέλη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λαζάρο για την παρουσίασή του και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έθεσε αυτή την έκθεση και υπό το φω του τέλους τη επόμενης προγραμματική περίοδου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο κ. Γκάιερ πολύ σωστά είπε ότι παρόλα τα θετικά ε, που λέει η έκθεση, η έκθεση πραγματικά δεν είναι πολύ αρνητική για την ε, Κομισιόν, παρόλα αυτά ε, υποδεικνύει συγκεκριμένε αδυναμίε. Δύο από αυτέ είναι εξή, όπω είπε ο κ. Γκάιερ. Πρώτον, το 38, στο 38% των περιπτώσεων ε, είχαμε ε, χαμηλή βεβαιότητα ότι τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση των κρατών μελών λειτουργούν σωστά μετά τις διορθώσεις. Και δεύτερον, δεύτερη αδυναμία, η οι διαδικασίες ε, για τη βελτίωση των συστημάτων αργούν. Παίρνουν πολύ χρόνο. Γνωρίζετε όμως ότι εργαζόμαστε επί αυτού εδώ και πολύ καιρό. Μην ξεχνάμε ότι η έκθεση αναφέρει στην περίοδο 2000-2006. Από τότε και μετά έχουμε καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουμε επιφέρει πολλές βελτιώσεις. Για παράδειγμα, εφαρμογή του προγράμματος του 2008 και οι επιπτώσει αυτού δεν φαίνονται στην έκθεση, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα, όπω ελέγχθη, να κάνουμε πρόσθετες διορθώσεις τη στιγμή της εκαθάριση του κλεισίματος και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη διαδικασία εκαθάριση των προγραμμάτων της τρέχουσα περίοδου και με τον νέο κανονισμό με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μάλλον, έχουμε πλέον περισσότερες δυνατότητες να παρέμβουμε εμείς ως Κομισιόν ε, και να επιφέρουμε διορθώσεις. Για παράδειγμα, διακοπή και αναστολή. Ε, δεν το βάζουμε κάτω. Κοιτάξτε την ετήσια έκδοση ε, δράσης 2011. Ε, έχουμε επιφυλάξεις σε το στο 1 τρίτο περίπου του συνόλου των προγραμμάτων. Και για αυτά τα προγράμματα προβαίνουμε σε πληρωμές μόνο όταν ικανοποιηθούμε με τη, από τη διόρθωση των αδυναμιών που έχουμε εντοπίσει. Αυτά για ό,τι αφορά την έκθεση. Τώρα, ο κ. Λαζάρου είπε κάτι πολύ ε, σημαντικό. Μίλησε για τη δυνατότητα αντικατάστασης μη επιλέξιμων δαπανών. Ο ισχύων κανονισμό επιτρέπει αυτή την αντικατάσταση ακόμα και αν εντοπίστηκαν οι αδυναμίες αυτές από, από, τον, εθνικ, από τον ε, από ευρωπαϊκό έλεγχο και συμφωνήσει το κράτος μέλος. Και αυτό είναι πρόβλημα. Η δική μας θέση είναι σαφής. Πρώτον, αν το κράτος μέλος εντοπίσει την αδυναμία, τη μη επιλέξιμη δαπάνη, τότε θα ε- πρέπει να έχει τη δυνατότητα να την αντικαταστήσει. Γιατί αλλιώ δεν δίνεται κίνητρο στο κράτο μέλο, στα κράτη-μέλη, να εντοπίζουν τέτοιου είδου αδυναμίε. Αλλά αν η αδυναμία δεν εντοπιστεί από το κράτο μέλος, αλλά από έναν έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντικατάσταση. Θα πρέπει να επιβάλλεται καθαρή διόρθωση, επιστροφή των ποσών. Και αυτό έχουμε προτείνει για τη νέα προγραμματική περίοδο. Και βασιζόμαστε στην νομοθετική αρχή. Και όταν λέω νομοθετική αρχή, προφανώς εννοώ ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρότασή μας θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο δίδαγμα που μπορούμε να εξάγουμε. Και υπάρχει και ένα δεύτερο. Που επίσης θα θέλαμε να βασιστούμε στη βοήθειά σας. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η ελέγχουσα ελεκτική αρχή ε, είναι υποχρεωμένη να ελέγχει με μεθόδου στατιστική δημοκρατοληψία. Αυτό για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, η στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, ε, για να διαθέτουμε μια ε, βάση, σταθερή βάση για τα συμπεράσματα και προκειμένου να εφαρμόσουμε μετά διορθώσει. Αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Όμως τι συμβαίνει τώρα. Το Συμβούλιο έβαλε μια αναφορά ξανά στο κείμενο συμβασμού σε μη στατιστική δειγματοληψία. Αν αυτό περάσει, οι ελεγκτικές αρχές θα, ε, θα δίνουν λιγότερη βεβαιότητα για τις αδυναμίες και θα γίνει πιο δύσκολο να εφαρμόσουμε τις διορθώσεις. Αυτό θα αποτελέσει μάλιστα μια υπαναχώρηση σε σχέση με τα στάνταρ που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή. Συνεπώ και εκεί θα ήθελα τη βοήθειά σας. Θα τελειώσω εδώ και ξανά ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο και τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. There is another opportunity. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντίφα. Καλό είναι να δώσουμε και στους συναδέλφους το λόγο για να μπορέσουν να θέσουν ερωτήματα. Η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα έχω. Το πρώτο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Είπατε ότι όταν διαπιστώνεται ένα λάθος ή κάποια προβληματικές έτσι, καταστάσεις, σταματάουν οι πληρωμές ή δεν γίνονται πλήρως οι πληρωμές. Μπορείτε να μας πείτε περίπου πόσο υψηλός είναι αυτός ο όγκος των παύσεων, δηλαδή των πληρωμών. Έτσι, χοντρικά. Δεν χρειάζεται να μας πείτε και τα δεκαδικά, αλλά καλό θα ήταν να, να δούμε τι τελικά σταματά από πληρωμές. Που πολιτικά δηλαδή θέλουμε να δώσουμε, αλλά λόγω των λαθών δεν δίνονται. Και δεύτερον, ε, θα μπορούσε να το απαντήσει η Κομισιόν ή ο εισηγητή δεν ξέρω, αλλά ε, στην, ε, στα όσα είπε το ελεκτικό συνέδριο μιλούμε για ποσοστό λαθών. Εγώ δεν είμαι τακτικά εδώ, οπότε ήθελα να μου πείτε αυτός ο όρος, ο ποσοστό λαθών, έχει να κάνει και με τη διαφθορά ή μιλούμε μόνο για λάθη, καθαρά λάθη. η κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, ευχαριστώ και τον ε, ε, εκπρόσωπο της, ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Κομισιόν. Είμαι της άποψης ότι η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική. Και μάλιστα σήμερα, κυρίως σήμερα και στην φάση που περνάμε. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε πολύ εντατικά με αυτή. Κανένας από εμάς δεν ε, θεωρεί ότι η ε, ε, πολιτική συνοχή είναι πολιτική δεύτερη κατηγορία. Είναι από τι πιο σημαντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να την προωθήσουμε. Σε σχέση λοιπόν με αυτό, θέλω να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Σε σχέση με την, τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε, κάνουμε, βρισκόμαστε στη φάση της διόρθωσης των διαφόρων λαθών, αλλά μιλούμε πάντα για τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτό όμως δεν εξηγείται, γιατί ένας ε, φορολογούμενος, ένας Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε εμείς μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι τώρα εμείς ζητούμε από την Κομισιόν ή της δίνουμε την εντολή να μας δώσει δεδομένα, ε, δηλαδή οικονομικές διορθώσεις που αφορούν στο έτος 2000-2006. Σήμερα Βεβαίω γνωρίζω ότι οι διαδικασίε είναι μακροσκελείς και κρατούν πολύ. Αυτό είναι σαφές. Αλλά θέλω να πω ότι για έναν φυσιολογικό πολίτη είναι τελείω ακατανόητο αυτό που γίνεται εδώ. Και γι' αυτό ακριβώ θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Στο μέλλον πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις μπορούν να μειωθούν. Είναι ένα ερώτημα για το μέλλον που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και επίσης να πω το εξής. Πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε πιο γρήγορα το πώς γίνονται οι διορθώσεις, εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα προβλήματα. Και κλείνοντας να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που ο εισηγητής ασχολήθηκε με τον συνολικό λογιστικό έλεγχο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα ο, ο έλεγχος αυτός ο λογιστικός ε, τη χάνει θετική ανταπόκριση από την έκθεση. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό γιατί αλλιώς θα δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα αν δεν έχουμε σαφείς και ενιαίους ε, κανόνες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Τσέσκοβα. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να πω απλώς ότι η παρούσα κρίση στα κράτη-μέλη έχει να κάνει και με την άρνηση των κρατών μελών για τα διορθωτικά ταμεία. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να το πούμε και να το συζητήσουμε ξεχωριστά. Για το ποιες δηλαδή είναι, ποια είναι τα δείγματα ή τα μαθήματα που μπορούμε να εξάγουμε από τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό των ε, ελεγχθέντων ποσών, των επιτόπου ελεγχθέντων ποσών από το ελεγχτικό συνέδριο. Περίπου 19% ε, είναι το ελεγμένο ποσοστό αυτό στη Γερμανία. Δηλαδή το 81% δεν ελέγχεται. Ε, υπάρχουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία και ναι που μπορώ να τα βρω. Επίσης, για το, εγώ ήμουν, εκπρόσωπ, ήμουν ε, εισηγήτρια για το 2011. Πραγματικά έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο ελεγχτικό συνέδριο. Ακούσατε όλα μας τα σχόλια και Μιλούμε για θέματα οικονομικών διορθώσεων που πλέον είναι πιο λίγες. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να πούμε πόσες είναι αυτές οι δηλώσεις των κρατών μελών που όντως είναι αληθείς, που είναι σωστές. Η Κομισιόν πόσες έχει ελέγξει και πόσες θεώρησε έγκυρες και σωστές και για τις, για τις διορθώσεις η κυρία Τσέσκοβα έχει δίκιο. Από το 2007 μέχρι το 2013 ο κανονισμός για, τον, για τα θερθωτικά ταμεία έχει τύχει ριζικής αναδιάρθρωσης. Οπότε δεν, τα όσα βλέπονται εκεί δεν ε, συνάδουν απόλυτα και με τα, ποσά που τελικά θα, θα διατεθούν. Έχουμε κάποια ελπίδα ότι τα χρήματα που θα ε, δοθούν όντως θα υπάρξουν ή απλώς θα διατηρήσουμε έτσι μία θεωρητική ιδέα και η επόμενη γενιά κοινοβουλευτικών θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν το, αν το δίκαιο δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, τι νόημα έχει να το προβλέπουμε. Πρέπει να πω ότι έχω δει τις ε, τροπολογίες ε, του ε, για τα διευθυντικά ταμεία και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές αλλαγές για την υποβολή των εκθέσεων, για τον, ε, την υποχρέωση των ελέγχων. Αν έρθουν όντως αυτά ε, προς εφαρμογή, θα μπορούμε πραγματικά να... Ό,τι ξέραμε μπορούμε να το ξεχάσουμε. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι ε, καλό είναι να μην υπάρχουν ε, έλεγχοι κτλ. για να ε, βελτιώσουμε και την γραφειοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έτσι θα, μπουν πολύ, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα κονδύλια από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συντονιστούμε και εδώ στην Επιτροπή μα για το τι θα κάνουμε με τον κανονισμό για τα διευθυντικά ταμεία και πώ θα ξεκαθαρίσουμε στου συναδέλφου ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια πράγματα ή κάποια από τι προτάσει τη Κομισιόν πρέπει να εγκριθούν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γκρέσλε. Αυτά λοιπόν ήταν τα ερωτήματα από τα μέλη της Επιτροπής. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντέφα να απαντήσει. Παρακαλώ. Βεβαίω, Πρόεδρε. Πρώτο σημείο της κυρίας Βάιλερ. Πόσο, ισχυρή είναι, πόσο ισχυρός είναι ο αντίκτυπος ε, της, ε, της πάυσης των πληρωμών. Έναν αριθμό μπορώ να σας πω για την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο βέβαια και που αφορά την παρούσα περίοδο. Είχαμε 3,5 δισεκατομμύρια πληρωμές, 3,5 δις ευρώ, τα οποία μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε εάν βεβαίως δεν ε, διακόπτονται τα προγράμματα. Αυτή είναι η κατώτατη, ο κατώτατος υπολογισμός, γιατί πολλοί δεν μας στέλνουν καν στατιστικά ή, ε, χρήματα, ή ε, στοιχεία γιατί ξέρουν ότι δεν θα πληρώσουμε. Οπότε, εντάξει, είναι σχετικό λίγο το ποσό που έχουμε. Το ποσοστό λάθους περιλαμβάνει το σύνολο των παρατυπιών, όχι μόνο λάθη, όχι μόνο διαφθορά, όλα μαζί, ούτε όχι μόνο απάτη, όλα μαζί. για το θέμα της πληροφόρησης για τις διορθώσεις. Η μόνη πηγή δεν είναι προφανώς η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο εξετάζει δείγματα και σε βάθος. Σε βάθος κάθε δείγμα. Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει περισσότερο πρόσφατη πληροφόρηση, όχι όμως τόσο λεπτομερή, μπορεί να τον παραπέμψουμε στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας. Εκεί κανείς μπορεί να βρει πληροφορίες για τον αριθμό των διορθώσεων και τα ποσά που αντιστοιχούν. Ε, Κυρία Γκρέσλε, πόσο μεγάλο είναι το ποσό των συναλλαγών που όντως ελέγχονται. Αν δείτε τι μα έχουν δηλώσει οι ελεκτικέ αρχές των κρατών μελών για την περίοδο αναφοράς ε, για, ε, για την ετήσια έκθεση 2011 θα δείτε ένα αριθμό ικανοποιητικό 35% Ειδικά αν έχετε υπόψη σας ότι αυτό, αυτά είναι αντιπροσωπευτικά, αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. Ε, νομίζω ότι θα έχετε έτσι μια γενική ιδέα καλή. Δεύτερο ερώτημα πόσες ε, ελεγκτικές αρχές είναι αξιόπιστες, αξιόπιστες περίπου τα 2 τρίτα. Έτσι, χοντρικά. Και τρίτο σημείο που ρωτήσατε, τι γίνεται με τις διορθώσεις. Αν όντως είναι, έχουν επιρροή σε εμάς. Όταν γίνει μία ε, όταν, από τη στιγμή που αρχίζει να ισχύει μια διόρθωση, με την συμφωνία βεβαίω του κρατου μέλους, τότε από την επόμενη, ε, ε, βγαίνει το ποσό από την επόμενη πληρωμή. Δεν περιμένουμε δηλαδή μέχρι, να, μέχρι το τέλος, γίνεται άμεσα α πούμε από την επόμενη πληρωμή γίνεται ο υπολογισμό. Ε, πρόεδρε, ελπίζω ότι έχω απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνοντας, Κύριε Λαζάρου, έχετε να προσθέσετε κάτι πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκάιαρ. Θέλετε μήπως και πάλι το λόγο, θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια των Ευρωβουλευτών. No, uh, thank you, Chair. Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ε, τίποτε άλλο να πω, εκτός αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις προς εμένα ειδικά. Ο κύριος Γκάιερ. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο. Η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αφορά μια περίοδο που έχει κλείσει. Την περίοδο δηλαδή μέχρι το 2006. Όπου ερευνήθηκε το αν όντω από τα κράτη-μέλη λαμβάνουμε, ε, γίνεται μάλλον ένας ε, ικανοποιητικό έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν μπορούσε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όταν διορθώνονται αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, πόσο γρήγορα διορθώνονται, πόσο γρήγορα τη δουν τα μελη στις προτάσεις της Κομισιόν για βελτίωση. Και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 2008 το πρόγραμμα δράσης του 2008 έχει όντως ε, συμπεριλάβει πάρα πολλά σημεία, έχει ε, ασχοληθεί με αρκετά από αυτά, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το πρόγραμμα δράσης. Ε, αν αυτό θα καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα με σχετικά με τις ελλείψεις που έχει σημειώσει το ελληνικό Συνέδριο για αυτή την περίοδο. Βεβαίως, θα μπορούσαμε εν τω μεταξύ να μιλούμε για μια αρκετά ικανοποιητική περίοδο μέσα στην οποία λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και μιλάω για αυτό που είπε η κυρία Τσέσκοβα. Ευτυχώς Και τώρα μιλάω για την έκθεση της ε, DigiRegio, με την οποία ασχολήθηκα ως εισηγητής για την ε, απαλλαγή της Κομισιόν, ότι η κριτική μας λειτουργεί. Η Κομισιόν δηλαδή ε, παρεμβαίνει πολύ πιο άμεσα για την αναστολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων όταν διαπιστώνει λάθη στα κρατη Και αυτό είναι κάτι που το έχει ζητήσει πολλές φορές η Επιτροπή μας. Να μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει, όταν τα λάθη είναι προφανή, να πηγαίνουμε κατευθείαν σε διόρθωση, γιατί το λάθος αυτό, γιατί το, το πιο εύκολος τρόπος να διορθώσουμε το λάθος είναι πριν δοθούν τα χρήματα, στο, μόλις το διαπιστώσουμε στο σύστημα. Γιατί έτσι μετά δεν θα υπάρξουν και λανθασμένες πληρωμές. Και τελικά αυτό θέλουμε. Και αυτό είναι το καλό νέο για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ότι η πίεση δηλαδή που ασκείται από την Επιτροπή μας προς την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία που έχει ε, πιο έγκαιρα, ε, δηλαδή την πάυση πληρώμων προς τα κράτη-μέλη, ότι όντως αυτό έχει τελικά αποτελέσματα. και είναι απαραίτητα τα κράτη-μέλη να δρουν έγκαιρα. διαβάζοντα αυτή την ετήσια έκθεση είδα ότι μόνο ότι και η Τσεχία μεταξύ άλλων ε, επηρεάστηκε πολύ από την ε, ε, πάυση πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπήρξε από την αρχή διαπίστωση του προβλήματος στην Τσεχία. Και ακριβώς λόγω της πίεσης της ε, Κομισιόν η Τσεχία πρέπει να διορθώσει το σύστημα ελέγχου της. Και αυτό γίνεται πιο γρήγορα πια. Αυτό σημαίνει άμεση απάντηση, ανταπόκριση σε ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Όντω η έκθεση δίνει σημαντικές, ε, σημαντικές προτάσεις και για το μέλλον. Ε, Βεβαίω από τα εισαγωγικά σχολεία του συναδέλφου Γκάιερ φαίνεται ότι η Κομισιόν δραστηριοποιήθηκε και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου η εισηγήτρια η κυρία Γκρέσλε είναι παρούσα. Προσπαθήσαμε λοιπόν οι οικονομικές διορθώσεις να παραμείνουν ε, στα πλαίσια του ε, δημοσιονομικού κανονισμού και ε, προτείνω το θέμα αυτό να το διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξη, ανεξάρτητα από το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα σε σχέση με την έκθεση Γκάιερ που έχει υποβληθεί για την έκθεση του Ελεκτικού Συναδρίου. Ε, ξέρετε ποιες είναι οι προθεσμίες. Τροπολογίες λοιπόν μέχρι τις 12 Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον κύριο Λαζάρου, τον κύριο Ντεφά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κλείνουμε το σημείο αυτό. Οπότε φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. μετά ε, αύριο θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στη συνεδρία των συντονιστών.